Καλησπέρα σας, κυρίες ε, και κύριοι. Ξεκινήσουμε την ετήσια διάλεξη της ε, ΣΤΟΑ, που φέτος έχει τίτλο «Η βιωσιμότητα της αηφορίας. Πώς η της αηφοριας πως η οικονομια θα εργαστεί για το περιβάλλον». Καλωσορίζω λοιπόν το κοινό μας εδώ πέρα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω εξηγώντας λίγο το τι είναι η ΣΤΟΑ. Η ΣΤΟΑ, η αξιολόγηση επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών, υπάρχει εδώ και 26 χρόνια. Στόχο έχει να αξιολογεί τις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες και να εξετάζει τις μακροπρόθεσμες επιλογές που έχουμε, κάτω που είναι χρήσιμο για τι πολιτικέ αποφάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα επιστημονικά στοιχεία χρειάζονται για να μπορέσουμε να λάβουμε τι σωστέ αποφάσει καθώ αυτέ επηρεάζουν πάρα πολύ στο μέσο πολιτική στόχο μας είναι να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ των επιστημόνων, των πολιτικών και του κοινού. Αυτό γίνεται με το να ενθαρρύνεται ο διάλογο. Η αιτήσια αυτή διάλεξη είναι η κορονίδα της δραστηριότητάς μας και δίνει ευκαιρία στους ευρωβουλευτές, στους επιστήμονες και το ευρύ κοινό να έρθουν σε επαφή με εμφανείς προσωπικότητες, επιστήμονες, επιχειρηματίες που μιλάνε για αντικείμενα που μας απασχολούν ιδιαίτερα. Η κλιματική αλλαγή, βιωσιμότητα, η κοινωνία της πληροφορίας, ιατρική έρευνα, αλλά και βεβαίως ανακαλύψεις ε, στην ε, βασική έρευνα. Έχουμε διερμηνία σήμερα σε 11 διαφορετικές γλώσσες και μεταδίδεται η συνεδρίαση στο διαδίκτυο, οπότε τα πράγματα που θα πούμε δεν θα μείνουν μόνο εντός αίθουσας. Το φετινό θέμα βεβαίω αφορά το πώς θα συμβιβαστεί η, οικονομική, η περιβαλλοντική εφορία και η οικονομική ανταγωνιστικότητα. Πώς θα τα ισορροπήσουμε αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Μήπως είναι ε, προτεραιότητες που αντιφάσκουν ή όχι. Είναι πάρα πολύ επίκαιρα τα ζητήματα αυτά. Η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στη Βαρσοβία. Και υπάρχουν πολλές συζητήσεις για την ε, αυξημένη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων όπως ο τυφώνας στις ε, Φιλιππίνες και το αν μπορούν να συνδεθούν με την κλιματική αλλαγή στοιχεία που αφορούν την ανθρώπινη επίδραση στην κλιματική αλλαγή συσσωρεύονται και επιβεβαιώθηκαν και από την τελευταία αξιολόγηση του διακυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή του IPCC. Σε μια έκθεση η παρουσιάστηκε στο κοινοβουλίο μας την προηγούμενη εβδομάδα. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να επιδείξει πως υπάρχει μια εναλλακτική πιο αηφόρος πορεία. Παραδείγματο χάρη, παίζουμε βασικό ρόλο στις προσπάθειες αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, ε, καλύτερης χρήσης ε, των πόρων του ύδατος. Επίσης σημαντικά βήματα έχουμε κάνει για να μετασχηματιστεί το ενεργειακό μας σύστημα όσον αφορά τις ανανεώσιμες υγείας ενέργειας, την αποτελεσματική χρήση ενέργειας και τη μείωση των ε, αερίων του θερμοκουπίου. Βεβαίως αυτό σημαίνει μεγάλο κόστος, αλλά είναι και ευκαιρία για καινοτομία, για καθαρή τεχνολογία και για κάποια δημιουργία θέσεων εργασία. Η πράσινη οικονομία είναι στη βάση της στρατηγικής του 2020 και στόχο έχει να επιτύχουμε έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη του 2020 ε, μετρήσιμη με κάποιους βασικούς δείκτες όπως παραδείγματο χάρη έργα και ανάπτυξη, απασχόληση, κλιματική αλλαγή ενέργεια και κοινωνική συμπερίληψη και θα συζητήσουμε βέβαια σε αυτή την ιδέα αργότερα. Όμως η οικονομική κρίση και η έλλειψη φιλοδοξίας στην σχετική πολιτική είναι παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε απογοητευτικά αποτελέσματα. Συζητάμε σήμερα που πολλά καράτη πλήττονται ακόμα από την οικονομική κρίση και αυτό έχει δραματικές συνέπειες για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Κάποιες κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν υψηλά δημόσια χρέη, η ανεργία ιδιαίτερα των νέων είναι ενισχυτική και δεν υπάρχουν πολλές ε, επενδύσεις ε, στην ε, οικονομική ανάκαμψη. Οπότε έχουμε πολλωμένη συζήτηση. Κάποιοι αρνούνται την κλιματική αλλαγή παρά τα επιστημονικά δεδομένα. Η οικονομική πολιτική επίσης θεωρείται πως, και, πως είναι αναποτελεσματική και δεν είναι φιλική προς τη βιομηχανία και βεβαίως ε, μειώνονται και οι περιβαλλοντικές ε, και κοινωνικές ε, προδιαγραφές. Στο πλαίσιο αυτού του διλήμματος έχει η Ευρώπη την πολυτέλεια να κοιτάει βράχη πρόθεσμα τις προκλήσεις αυτές. Πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τους εταίρους μας προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα κάποιους εκλεκτούς ομιλητές για να δούμε κάποια από αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω στην ετήσια αυτή διάλεξη και όσους βεβαίως συμμετέχουν από απόσταση. Βεβαίω, αυτό ωφελεί το περιβάλλον. Οπότε κατά μία έννοια ταιριάζει με το θέμα μας. Άνθρωποι που θα έρχονταν στις Βρυξέλλες μπορούν να δουν τη διάλεξη αυτή στην ιστοσελίδα μας. Και έτσι μειώνει το αντίκτυπο στο περιβάλλον. Όσοι βλέπουν δε το ε, site μπορούν να στείλουν μηνύματα μέσω κάποιων hashtags, το hashtag δηλαδή στο 2013 στο Twitter. Τώρα, να σας παρουσιάσω τους ομιλητές μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Βλάσακ, τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον αρμόδιο για τη ΣΤΟΑ, για το μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, καθώς δυστυχώς είχε κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Θα επισημάνει ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συνεχίσουμε προς μια πορεία περιβαλλοντικής αηφορίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο πρώτος μας ομιλητής ε, θα είναι ο καθηγητής ε, Ισμαήλ Σεραγγελντίν, διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Ε, θα μιλήσει βεβαίως για το περιβάλλον και την κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη, θα αναπτύξει νέους τρόπους σκέψης, μέτρα και πολιτικές. Ο Ισμαήλ Σεραγγελντίν θεωρεί πως χρειάζεται μια πιο βαθιά αλλαγή στην οικονομική ανάλυση και στους δείκτες που χρειάζεται πολιτικής. Θα αναφερθεί στην εφορία ως ευκαιρία. Μετά τον ε, κύριο Σεραγγελδίν θα ακούσουμε ένα μήνυμα του κυρίου Χακίμ, Ακίμ Στάινερ, εκτελεστικού διευθυντή του προγράμματος περιβάλλοντος ε, του ΟΗΕ και αναπληρωτή γενικού γραμματέα. Θα μιλήσει για την εφορία και τις ανανεώσιμες φυγές ενέργειας. Το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΙΕ στοχεύει να βοηθήσει την αηφορία και την κοινωνική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Μόνικα Κίρχερ, διευθύνουσα σύμβουλος της Infineon Technologies Austria ΑΕ η οποία θα μας μιλήσει για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις ε, μεταφορές και το περιβάλλον. Η εταιρεία της ε, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική εφορία και βεβαίως ε, έχουν βραβευτεί πολλά και γι' αυτό. Η Μόνικα Κίρχερ και η διεθνή ομάδα της δημιουργούν παγκόσμιες τάσεις και στόχο έχουν την υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών με τα καινοτόμα προϊόντα τους. Μετά θα ακούσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Hans Brüning, εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Θα αναφερθεί στο ζήτημα της διαχείρισης της αλλαγής ε, με τη χρήση τεχνολογικών στοιχείων και κοινωνικών εταίρων. Αυτό το οποίο λέμε κοινωνιοτεχνικά συστήματα. Τέλος, θα ακούσουμε την ε, καθηγήτρια Αν Γκλόβερ, επικεφαλής ε, επιστημονική σύμβουλο του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Παλ Ρούμπιχ, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Ο Μάλκομ Χάρμπορ, επίσης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας ε, και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς, θα διευθύνει τη συζήτηση. Έχει μεγάλη εμπειρία, καθώς ε, ήταν ε, ο συντονιστής της ε, περισσότερες συζητήσεις τα τελευταία 4-5 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Τον λόγο έχει ο Μάλκομ Χάρμπορ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αντώνιο. Ευχαριστώ και σε σένα αλλά και, την, και σένα και την ομάδα που συγκέντρωσες ένα εξαιρετικό σύνολο ανθρώπων σήμερα το απόγευμα. Απλώ εγώ συντονιστή να κάνω κάποια σχόλια, να πω ότι ε, θα προσέχω το χρόνο μιλίας για να έχετε και χρόνο για ερωτήσεις ε, στο τέλος. Ε, έτσι λοιπόν, να χρειαστεί να σας κάνω να μιλήσετε πιο γρήγορα, θα χτυπάω εδώ το σφυράκι μου. Υπάρχουν και κάποιες διαφάνειες, έτσι λοιπόν μπορείτε να τις βρείτε έξω από την αίθουσα, αλλά θα υπάρχουν και στην οθόνη οι διαφάνειες αυτές. Το άλλο σημαντικό είναι ότι ήθελα να σας ενθαρρύνω να σκεφτείτε ερωτήσεις που θέλετε να θέσετε. Όταν εγώ προεδρεύω της Επιτροπής, ξέρω ποιος είναι ο καθένας. Σήμερα έχουμε μεγάλο κρατήριο. Θα σας δώσουμε και κάποια έντυπα για ερωτήσεις που θα κυκλοφορούν και κατόπιν θα τα συλλέξουμε και θα τα συγκεντρώσουμε εδώ στον οργανωτή. Έτσι λοιπόν σας ενθαρρύνουμε να θέσετε κάποιες ερωτήσεις και σας παρακαλώ να σημειώσετε και τις ερωτήσεις σας. Την περασμένη φορά έδωσα το λόγο σε κάποιον και ξέχασε τι ήθελε να ρωτήσει. Έτσι λοιπόν, σας παρακαλώ, αν ε, θέλω να παρουσιάσω την ερώτησή σας ερωτικά, θα αναφερθώ και στο σχετικό έγγραφο. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ερωτήσεις και στο Twitter. Και φαντάζομαι ότι όλοι τώρα θα ασχολείστε με το Twitter σχετικά με την εκδήλωση αυτή. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε ένα μεγάλο επίπεδο αλληλεπίδρασης. Και κάτι ακόμη που θα ήθελα να πω, κυρίως σε όσους μας παρακολουθούν από το ίντερνετ, ε, θα έχουμε και διερμηνία σε 11 γλώσσες σήμερα. Και χάρη στα θαύματα της τεχνολογίας μπορείτε να ακούσετε και τη γλώσσα της επιλογής σας στο διαδίκτυο μέσω web streaming. Εργάζονται σκληρά διερμηνείς εδώ στις καμπίνες. Να σας πω ότι θα έχουμε αγγλικά, τσεχικά, ουγγρικά, πορτογαλικά, ιταλικά, γερμανικά γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, σουηδικά, ελληνικά. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Μπορείτε λοιπόν να ακούσετε αυτές τις γλώσσες. Αυτά σχετικά με το επίσημο μέρος. Καταρχήν θα δούμε ένα μήνυμα στο βίντεο από τον Αντιπρόεδρο Βλάσακ Έχουμε ήχο, παρακαλώ. Δεν υπάρχει ήχος. What happened to the sound? Τι συνέβη με τον ήχο. Να σας δώσω λίγο χρόνο για να το λύσετε το πρόβλημα. Θα πρέπει να λύσουμε τα τεχνολογικά προβλήματα. Είχαμε και προηγουμένως ένα μήνυμα πώς ε, μπορούμε να πετύχουμε την ε, βιωσιμότητα, πώς μπορούμε να ανατρέψουμε τις αρνητικές περιβαλλοντικές αλλαγές. κύριε και κύριοι, ως ε, Αντιπρόεδρος υπεύθυνο για την αξιολόγηση επιστημονικών και τεχνικών επιλογών, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ετήσια διάλεξη της ΤΟΑ. Το παγκόσμιο περιβάλλον ε, παραμένει ένα ζήτημα που συζητείται τα μάλλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την περασμένη εβδομάδα η ΣΤΟΑ υλοποίησε ένα εργαστήριο για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην ε, έκθεση IPPC 2013. Από τη συζήτηση αυτή προέκυψε μια κυρία ερώτηση πώς μπορούμε να πετύχουμε τη βιωσιμότητα Πώς μπορούμε να ανατρέψουμε τις αρνητικές περιβαλλοντικές αλλαγές που τονίζονται σε αυτή την έκθεση της IPCC ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής μας και την παγκόσμια οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί η σημερινή συζήτηση θα μπορούσε να μας δώσει τη σκοπούμενη απάντηση. Επομένως, με μεγάλη ικανοποίηση καλωσορίζω τους σημερινούς ομιλητές, ε, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες, αξιόλογους που θα μας ε, παρουσιάσουν τις απόψεις τους για το πώς το αν εργαστούμε προς ε, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, νέες αγορές και νέες βιομηχανίες και νέους κλάδους. Εγώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρώ ότι θα πρέπει να διατυπωθεί αυτό το κύριο ερώτημα. Η δημόσια υποστηρίξη της έρευνας και της καινοτομίας ποια μορφή πρέπει να πάρει προκειμένου να συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στην αηφοροανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ζωτικό την επιδίωξή μας να μειώσουμε τις αρνητικές περιβαλλοντικές αλλαγές, να μην κλείνουμε τα μάτια μας σε δύο τεινά. Καταρχήν τον οικονομικό ξορθολογισμό και δεύτερον τη σημασία της βιομηχανίας ε, και της ε, δραστηριότητας ε, που κινείται με γνώμονα την καινοτομία. Το, η σημασία της, του οικονομικού εξορθολογισμού είναι σαφής όταν δούμε παραδείγματα δημοσίων επιδοτήσεων ε, στα φωτοβολταϊκά. Έχουμε ε, την ε, πρόθεση μάλλον ο οικονομικό έχει επισκιαστεί από την πρόθεση απλώς να πετύχουμε τους στόχους των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Αυτή, στο συγκεκριμένο τομέα έχει επεκταθεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό σε ένα αριθμό κρατών μελών και απειλούνται οι θέσεις ε, εργασίας ε, σε κάποιες ενεργοβόρες βιομηχανίας ε, λόγω αυξηνόμενων τιμών ενέργειας. Τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την άποψή μου με ένα άλλο παράδειγμα. Προέρχομαι από την Δυσική Δημοκρατία και μπορεί να μην σας εκπλήξει ότι αυτό το παράδειγμα αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Στον τομέα αυτό η έρευνα και η καινοτομία είναι αναγκαιότητα, απόλυτη αναγκαιότητα για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και για να σεβαστούμε τους στόχους εκπομπών της Ευρώπης. Τολμώ να πω ότι αυτή είναι επιλογή τη συμμερίζονται ευρέως πολλοί νομοθέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η βιομηχανία. Όμως, ενώ ε, μπορεί ενίοτε να αποκλίνουν οι απόψεις τους, είναι ελεύθερη επιλογή του κλάδου κυρίως ε, σε ποιους τομείς θα επικεντρώσουν την έρευνά τους. Εγώ ως εισηγητής στην Επιτροπή Μεταφορών ε, για το CARS 2020, για το σχετικό σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία, έχω στήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Είμαι βαθιά πεπισμένος ότι αν οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να περιορίσουν αυτή την ε, δυνατότητα επιλογής. Το αποτέλεσμα θα ήταν να ε, μειωθεί συνολικά η τεχνολογική πρόοδος καθώς και οι εκπομπές. Παραδείγματος χάρη, αν ε, κατευθύνουμε όλους τους παραγωγούς σε μια έρευνα των για τον μπροστινό τμήμα ε, του οχήματος, τότε περιορίζουμε την εστίασή του σε συγκεκριμένους τομείς, όπου περιορίζουμε του τους οικονομικούς ε, πόρους που θα μπορούσαν να εξελιχθούν αλλιώς και να χρησιμοποιηθούν και να επενδυθούν σε άλλους τομείς όπως θα ήταν τα λάστιχα, οι μηχανές, ε, τα τρένα ή τα αεροδρομική στο πίσω μέρος του οχήματο. Η άποψή μου, επομένως, είναι πάρα πολύ απλή και τη διαβιβάζω εδώ στο κοινό. Να αφήσουμε τους νομοθέτες να νομοθετήσουν σχετικά με τους στόχους και τους ερευνητές να ερευνούν. Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Μάλκομ Χάρμπορ, τον αντιπρόεδρο της ΤΟΑΣ και τον σημερινό συντονιστή της συζήτηση, να μου επιτρέψετε να δράξω αυτή τη στιγμή για να σας ευχαριστήσω όλους εσάς για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη διάλεξη. Η συμμετοχή σας ημέρα μας ε, δείχνει ότι ενδιαφέρεστε και για την καταπολέμηση της ενεργείας και για την προστασία του περιβάλλοντος και δικαίως ενδιαφέρεστε καθώς εδώ διακυβεύεται η ποιότητα της ζωής του καθένα μας. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Αντιπρόεδρο Λάσεκ για αυτό το μήνυμα και μπορούμε να ξεκινήσουμε την συζήτηση, να ακούσουμε τις ομιλίες των προσκεκλημένων μας. Είναι τιμή για μένα να ζητήσω από τον κύριο Σαραγγέλτη να διευθύντη της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας να μας μιλήσει. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που καταφέραμε να τον φέρουμε στις Βρυξέλλες. Είχε επισκεφθεί, τον είχα γνωρίσει μάλλον πριν 8 χρόνια στην Ιαπωνία. Είναι παγκοσμίω γνωστό, διάσημο επιστήμονα. Είναι μεγάλη τιμή για μα που ήρθατε. σα καλωσορίζω. Και σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, προετοιμάζεται τεχνικά η παρουσίαση μου αναρωτιέμαι αν μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες. Ναι, ωραία. Τώρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κυρίε και κύριοι, θέλω να σα μιλήσω για το περιβάλλον και την κοινωνική βιωσιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να την υλοποιήσουμε αυτήν μέσω νέα νοοτροπία και νέων μέτρων πολιτική. Αυτό είναι το περιεχόμενο της παρουσίασης μου. Θα κλείσω για δείκτες πέρα από το ΑΕΠ. Τα πρώτα βήματα που έχουν γίνει σας προς αυτή την κατεύθυνση. Με ποιον τρόπο μπορούμε να δούμε την βιωσιμότητα ως ευκαιρία. Με ποιον τρόπο αυτή μπορεί να συνεισφέρει στην ζωή των πολιτών ζητήματα που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα του θέματο και τέλο θα μιλήσουμε για το γιατί χρειάζεται να αναλάβουμε δράση τώρα και γιατί ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Α ξεκινήσουμε πρώτα από το ζήτημα του ΑΕΠ. Φαντάζομαι γνωρίζετε αυτά τα θέματα, αλλά έχουν ε, πολλοί οικονομολόγοι όπω ο κ. Στίγκλιτ εκφράσει ανησυχίε για τη χρήση αυτή του ΑΕΠ ω ε, τρόπο μέτρηση. Υπάρχουν άλλοι δείκτε, όπω για παράδειγμα το λεγόμενο Cross National Happiness ακαθάριστη εθνική ευτυχία, ας μπορούμε να τη μεταφράσουμε, είναι ένας δείκτης ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη, χωρίς όμως αυτή η χρήση του να εξαπλωθεί στον υπόλοιπο κόσμο. Στοιχεία για την Ευρώπη μπορείτε να δείτε σε αυτή τη διαφάνεια. Προσπαθούμε λοιπόν να κατατήσουμε εναλλακτικούς δείκτες ως προς το ΑΕΠ. Ίσως το Human Development Index, ο δείκτης ανθρώπινης ε, ανάπτυξης του ε, προγράμματος περιβάλλοντος του ΙΕ, να είναι ο πιο υποσχόμενο τέτοιο δείκτης. Επίσης είναι σημαντικό να μετρά κανείς την ανισότητα ε, στην κοινωνία, γιατί αυτό ουσιαστικά αναφέρεται στο κατά πόσο οι πολίτε ατομικά μπορούν να απολάβουν τις βελτιώσεις στην κοινωνία και διαπιστώνουμε αύξηση των ανισοτήτων. Για παράδειγμα το 2012 μειώθηκε κατά 12% αυτός ο δείκτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν λάβουμε υπόψη μας λοιπόν τις ανισότητες και στη σχετική κατάτηξη οι Ηνωμένε Πολιτείες κατέβηκαν 13 θέσεις. Επομένω, είναι σημαντικό. Ε, προσπαθώντας τώρα να κοιτάξουμε την πλευρά της οικολογικής βιωσιμότητας διαπιστώνουμε ότι η χρήση αυτού του δείκτη δεν είναι και τόσο χρήσιμη όπως το ίδιο συμβαίνει και με το ΑΕΠ ανακατακεφαλή. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ του δίκτυα αυτού και της οικολογικής, του οικολογικού αποτυπώματος. Τι σημαίνει αυτό. Ότι όσοι είναι πλουσιότεροι, οι κοινωνίε οι οποίε είναι πλουσιότερες έχουν μεγαλύτερο οικολογικό αποτύπωμα. Αυτό το γνωρίζαμε ήδη, αλλά έχει επιπτώσει για τι πολιτικέ μα επιλογέ. Με άλλα λόγια, κανένα από αυτού του δείκτε δεν μα βοηθά να ε, κατευθυνθούμε προ μια πιο ε, βιώσιμη οικονομία. Επομένω, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψη μα. Και ποια είναι τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για τους εθνικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο περιβάλλον. Και προσπαθήσαμε να πείσουμε τα Ηνωμένα Έθνη να λάβουν μια πρωτοβουλία έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνεται το περιβάλλον στην ε, ε, δημόσια λογιστική, στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη παρακολουθούν του λογαριασμού του. Γιατί. Αυτή τη στιγμή το να υπάρχει ένα δάσο σε μια χώρα μετρά μηδέν, δεν μετρά. Εάν αρχίσει η υλοτομία και καταστραφεί αυτό το δάσο, αυτό καταγράφεται ω θετικό Επομένω, είπαμε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται το περιβάλλον στην ε, δημοσιολογιστική και είπαμε ότι πρέπει να καταγράφονται τέτοιου τύπου επιπτώσει. Ποιε είναι οι επιπτώσει στο φυσικό περιβάλλον και σε δεύτερο στάδιο αυτές οι επιπτώσεις πώς επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού. Και τελικά ποιε είναι οι επιπτώσει στην οικονομική ανάπτυξη. Και τέλος, σε τρίτο επίπεδο, ε, φτάνουμε και σε μια ε, οικονομική επιμέτρηση του προβλήματος, μια ποσοτικοποίηση του με οικονομικούς όρους. Και συνδυάζοντας τους ε, συνήθεις λογαριασμούς ενός κράτους τον ισολογισμό του με αυτούς τους περιβαλλοντικούς οικολογικούς λογαριασμούς, μπορούμε να φτάσουμε στους λεγόμενους πράσινους λογαριασμούς. Ωστόσο, η συνήθις ε, δημοσιολογιστική παραμένει ο τρόπος με βάση τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις κατά κύριο λόγο παντού, σε όλες τις χώρες. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την Ηνωμένα Βασίλεια να προσπαθήσουμε να αποσυντικοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι περιβαλλοντικές ανησυχίες μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομία, εξοικονόμηση. Ε, διαπιστώνουμε εδώ στα αριστερά 22% ακαθαριστή εθνική επένδυση. Αν λάβουμε υπόψη μας τις αποσβέσεις φτάνουμε στο 12%, εάν λάβουμε υπόψη μας την επίπτωση στους φυσικούς πόρους φτάνουμε στο 5% και αν τελικά λάβουμε υπόψη μας και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αυτή η επένδυση είναι, οδηγεί σε μείον 2% στο, στο ΑΕΠ. Άρα αλλάζει τελείως η εικόνα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να πάμε πέρα από την περίπτωση του Μεξικού που μόλι είδαμε και να εφαρμόσουμε την ίδια μεθοδολογία σε όλε τι χώρε τη Λατινική Αμερική. Βλέπετε εδώ τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε υπόψη μα τη μία παράμετρο μετά την άλλη και δεν μα εκπλήσει καθόλου ότι τελικά αυτέ οι εξοικονομήσει ήταν ακριβώ το αντίθετο. Δεν, δεν, ε, ε, δίνουν ακριβώς την αντίθετη εικόνα από τη θετική εικόνα που μα έδιναν ε, τα οικονομικά στοιχεία από μόνα τους. ένας οικονομολόγος θα σας επισημάνει ότι αυτά τα στοιχεία, ε, αυτές οι καμπύλες έχουν την ίδια δομή. Όμως εδώ κρύβεται μια πολύ σημαντική διαφορά, μια ε, διαφορά της τάξης του 10%. Επομένω το ερώτημα είναι πόσο εξιόπιστη μπορεί να είναι αυτή η μεθοδολογία μέτρησης και αυτή η καμπύλη. επαναλάβαμε το ίδιο τρόπο μέτρησης για όλες τις χώρες του κόσμου. Και τι μας εντυπωσιάζει εδώ ως έβριμα. Ότι αν κοιτάξουμε στη δεκαετία του 80, θα διαπιστώσετε ότι η Ανατολική Ασία απογειώνεται ενώ στην υποσαχάρια Αφρική η καμπύλη καταραίει και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με την αντίληψη που έχουμε για την πραγματικότητα. Επομένως αυτή η μεθοδολογία, αυτές οι καμπύλες μετρούν κάτι πραγματικό, μετρούν την πραγματικότητα, κάτι που, που κρύβεται με τους συνήθεις οικονομικούς δείκτες. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και μας δείχνει πόσο απαραίτητο είναι να υιοθετηθεί αυτή η μεθοδολογία των πράσινων δημόσιων λογαριασμών είναι ένα σημαντικός δείκτης προκειμένου να μεταβούμε προς μια βιώσιμη αηφόρο οικονομία. Δηλαδή δεν αρκεί κανείς να μετρά μόνο τις επενδύσεις ως προς το ΑΕΠ. Αυτό μπορεί να κρύβει ε, άλλας πραγματικότητας. Με ποιον τρόπο λοιπόν μπορούμε να μεταβούμε προς την βιώσιμη ανάπτυξη. Σας δείχνω εδώ τον ορισμό της Επιτροπής Bratland, οποία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αυτή η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να συνεισφέρει στις μελλοντικέ γενναίε. Υπέροχο ορισμό, αλλά ανεφάρμοστο στην πράξη. Γιατί δεν μα λέει τι θα κάνουμε με αυτού, για παράδειγμα, που έχουν ήδη δύο αυτοκίνητα στην κατοχή του. Μα μιλάει για τι μελλοντικέ γενναίε. Τι θα πρέπει όμω να γίνει με τι σημερινέ. Το ερώτημα που κρύβεται πίσω από αυτά είναι ποιε είναι οι πραγματικέ ανάγκε ενό ανθρώπου. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε έναν άλλον ορισμό, πιο πρακτικό. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιες ε, ε, είναι οι διάφορε ε, σχέσεις μεταξύ τη βιωσιμότητα και του περιβάλλοντος, αλλά δεν ήταν πολύ πρακτικό αυτό. Επομένως θεωρήσαμε ότι πρέπει να δούμε την βιωσιμότητα ως ευκαιρία. Και ο ορισμό που δίνουμε είναι ότι η εφορία πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι μελλοντικέ γενναίε θα έχουν τι ίδιε, εάν όχι περισσότερε ευκαιρίε από αυτέ που έχουμε εμεί σήμερα. Με άλλα λόγια, λένε ότι οι μελλοντικέ γενιέ θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή του μεγαλύτερε δυνατότητε, μεγαλύτερε ε, ευχέρεια να δημιουργήσουν πλούτο κατά κεφαλή. Γυρνώντα λοιπόν στην οικονομική βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική βιωσιμότητα, διαπιστώνουμε ότι η οικονομική βιωσιμότητα αναφέρεται κυρίως στον πλούτο, στο κεφάλαιο που παράγεται από τον άνθρωπο, το, η οικονομική βιωσιμότητα αναφέρεται στους φυσικούς πόρους και στην κοινωνική βιωσιμότητα είναι ο συνδυασμός ε, του, του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού κεφαλαίου. Πρώτη διαφάνεια λοιπόν τα λεωφορεία είναι αυτό που θα ονομάζαμε παραδοσιακά έτσι, ανθρωπογενείς πόρους, ε, μετά σας έδειξα την, το δάσος φυσικό, φυσικό περιβάλλον και μετά έχουμε την κοινωνία, οι φωτογραφίες από τα σχολεία. Τι θέλουμε λοιπόν να μετρήσουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε μάλλον. Αυτά τα τέσσερα είδη κεφαλαίου, κατά κεφαλή, να αυξάνονται ή να παραμένουν ε, τα ίδια αποδεχόμαστε ότι η κατανομή μεταξύ αυτών των τεσσάρων εδών κεφαλαίου θα αλλάξει. Για παράδειγμα στη Ζάμπια όπου υπάρχει δυνατότητα εξόριξης χαλκού θα μειωθεί το φυσικό περιβάλλον, θα μειωθούν οι φυσικοί πόροι αλλά θα αυξηθούν οι κοινωνικοί πόροι γιατί τα έσοδα από αυτή την εξόριξη χαλκού θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση. Αλλά και στα τέσσερα είδη κεφαλαίου υπάρχουν όρια. Όρια στο πόσο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε προκειμένου να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε ε, πρακτικά να το εφαρμόσουμε αυτό. Ναι, τα καταφέραμε, το εφαρμόσαμε σε 130 χώρες και καταφέραμε να μετρήσουμε ε, τον πλούτο τους. Αυτό που ε, ξεκινήσαμε το 1995 με μια έκθεση που εξέδωσε η Παγκόσμια Τράπεζα παρακολουθώντας την περιβαλλοντική πρόοδο, Monitoring Environmental Progress και εδώ σας δείχνω κάποια από τα αποτελέσματα αυτής ε, ε, χωρίζουμε τις χώρες σε τρεις ομάδες, εκείνες που εξάγουν φυσικούς πόρους, εκείνες που είναι αναπτυσσόμενε και εκείνες οι οποίε ε, έχουν ήδη υψηλά εισοδήματα με μπλε είναι τα παραγόμενα αγαθά, το κόκκινο είναι το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και φυσική πόρη με κίτρινο. Κάναμε την ίδια διαδικασία για 100 χώρες το 1997 με την ίδια μεθοδολογία κάπως βελτιωμένη και διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στην κατανομή. Άρα, αυτό που διαπιστώνουμε είναι το 80% του, του πλούτου προέρχεται από το ανθρώπινο και το φυσικό κεφάλαιο. Επομένως, εκεί πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειες μας για την βιωσιμότητα. Δεν θα πρέπει λοιπόν η χρήση των φυσικών πόρων να υπονομεύει αυτά τα δύο είδη κεφαλαίου. Επαναλάβαμε την μελέτη για το Βέλγιο και την Αίγυπτο σε μεγαλύτερο βάθος. Αποτέλεσμα ήταν το βιβλίο Social Capital, κοινωνικό κεφάλαιο. Νομίζω ότι αυτό, αυτή η αρχή υπόσχεται πολλά, αλλά να γίνουν. Θα ήθελα τώρα να σα δείξω τον τρόπο με τον οποίο αυτέ οι πολιτικέ, αυτή η διαφορετική πολιτική θα βελτιώσει την ζωή, την ζωή των ίδιων των ανθρώπων θα, θα σταθώ μόνο στα σημαντικά θέματα. Το σημαντικό είναι η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων να μην ε, χειροτερεύει, να βελτιώνεται. Ας κοιτάξουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα το προσδόκιμο ζωής. Η καμπύλη εδώ ότι προφανώς ότι δεν είναι γραμμική και έχει αλλάξει η κύρτωσή της από το 60 μέχρι το 87. Ε, εδώ έχουμε το εισόδημα από 0 έως 20.000 ε, δολάρια κατά κεφαλή και το αντίστοιχο προσδόκιμο ζωής. Για την καλύτερη περίπτωση, το μεγαλύτερο εισόδημα, διαπιστώνεται ότι δεν αυξάνει και πάρα πολύ το προσδόκιμο ζωής. που είναι σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 80% του πληθυσμού βρίσκεται στα αριστερά της διοικημένης γραμμής, δηλαδή κάτω από 10.000 δολάρια κατά κεφάλι. Αυτό όμως που διαπιστώνουμε ότι είναι με τον ίδιο ε, με, με την ίδια ποσότητα πόρων αλλά με βελτιωμένη πολιτική καταφέρνουμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη βελτίωση γιατί, για παράδειγμα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιστημονικά εργαλεία για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των ε, ε, μητέρων, την υγεία τους, ε, να μειώσουμε τη μητρική θνησιμότητα, έχουμε καλύτερη ιατρική περίθελψη. Και θα διαπιστώνουμε ότι θα έπρεπε να αυξηθεί αν προσπαθούσαμε άλλο να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αυξάνοντας το εισόδημα θα έπρεπε να το οκταπλασιάσουμε. Το ίδιο αποτέλεσμα που μπορούμε να το έχουμε με, με βελτιω, βελτίωση της πολιτικής. Η απάντηση όμως που θα μου δώσετε είναι ναι, ωραία όλα αυτά, αλλά οι εποχές τις οποίες ζούμε είναι πολύ περίπλοκες και θα έλεγα σχεδόν χαοτικές. Πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά που λέτε στην πράξη σήμερα. Ε, θα έλεγα ότι μπορούμε και τώρα μόλις ξεκινάμε. Όταν κανείς βλέπει ένα κτίριο αρχιτεκτονικά ή την γεωμετρία ενός λουδιού μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ περίπλοκο, αλλά στην πραγματικότητα βασίζεται σε απλά δομικά υλικά. Όλα αυτά ο αριθμός στα πέταλα σε ένα λουλούδι, στα, στα φύλλα ή τα, σύννεφα ή ακόμα και οι πυραμίδες, όλα αυτά αν τα δει κανείς στο σύνολό τους είναι πάρα πολύ περίπλοκα, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούνται από πολύ πολύ μικρά στοιχεία, εύκολα να τα αντιληφθεί κανείς. Το ίδιο μπορούμε να διαπιστώσουμε και στα φράκτα. αρχικά τα φράκταλ, τα μορφοκλάσματα έγιναν διαδεδομένα, γιατί είναι, ε, έγιναν δημοφιλή μάλλον γιατί είναι όμορφες εικόνες. Αλλά στην πραγματικότητα εξηγούν με μαθηματικό τρόπο πολύ σημαντικά φυσικά φαινόμενα ή πολύ σημαντικά άλλα φαινόμενα όπως για παράδειγμα το, το χρηματιστήριο. Ωραία χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή για παράδειγμα για την εξήγηση της διακύμανσης των τιμών μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα αυτή την καπήλη η οποία φαίνεται πολύ περίπλοκη της διακίνησης σε ώρες, ημέρες, εβδομάδες, ό,τι και αν είναι και να την εξηγήσουμε. Για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές ε, ε, διαφορετική γεωμετρία, διαφορετική μεθοδολογία γεωμετρική από την παλιά. Όλα λοιπόν αυτά μας βοηθούν καλύτερα να καταλάβουμε πολύ διαφορετικά μεταξύ τους φαινόμενα, όπως για παράδειγμα τη δομή των υφάδων, το DNA, τη δομή των λουλουδιών ή ακόμα και τους, τους καρκίνους ή ακόμα και την οργανική ύλη ή τα νευρονικά δίκτυα. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα νοοτροπία, ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων και τώρα μόλις ξεκινούμε. Το ερώτημα λοιπόν στο οποίο έρχομαι, γιατί να αναλάβουμε δράση τώρα και γιατί να το κάνουμε αυτό στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτή η νέα νοοτροπία για την οποία σας μίλησα έρχεται σε μια στιγμή που αλλάζει εκφάθρον ο τρόπος σκέψης των οικονομολόγων και οι οικονομικές σχολές. σα είπα πριν τη θέση των Στίγκλιτς, των Σεν και σε σχέση με το ΑΕΠ, βραβευμένοι με τον Νόμπελ, ένας άλλος οικονομολόγος βραβευμένος με Νόμπελ, ο Κρούκμαν, ε, διαφωνεί πλήρως με τη σχολή του Σικάγο. Ο Στίγκλιτς ε, επιτέθηκε στο, στην ε, παγκοσμιοποίηση και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί Πρόσφατα έχουν δημοσιευτεί από σοβαρούς και διάσημους κονομολόγους βιβλία για την Ινδία, τρία βιβλία για την Ινδία. Με τους τίτλους που βλέπετε στις οθόνες. Και επίσης ο Άρβιν Παναγαρέτα δημοσίευσε ένα βιβλίο, εξέδωσε ένα βιβλίο με το τίτλο «Γιατί έχει σημασία η ανάπτυξη». Ο Σεν και ο Ντρέζε μας λένε ότι αν εξετάσουμε πιο προσεκτικά τον ρυθμό ανάπτυξης της Ινδίας θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι πραγματικός γιατί υπάρχουν τεράστιες ανισότητες και αντιθέσεις στην Ινδία. Ο ένας αναφέρεται στο κράτος πρόνοιας, ο άλλος αναφέρεται στις επενδύσεις ο πληθυσμός της Ινδίας θα αυξηθεί με κατά 100 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια και θα χρειαστεί αυτός ο πληθυσμός να τραφεί και να ζήσει με τους ίδιους φυσικούς πόρους. Πώς θα γίνει αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συζήτηση σε εξέλιξη και έχει έρθει πια η ώρα να αλλάξει η ορθόδοξη οικονομική σκέψη. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη. Είναι το, γνωστό ερώτημα του εάν το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Αν είμαστε ε, απεσιόδοξοι ή αισιόδοξοι στην προσέγγιση μας. Οι λαοί στην Ευρώπη ήδη δηλώνουν την αντίθεσή τους, διαδηλώνουν την αντίθεσή τους σε αυτές τις πολιτικές και ζητούν να αλλάξουν. Οι αλλαγές αυτές φυσικά δεν θα είναι εύκολες, θα πρέπει να αποδεχθούμε νέες τεχνικές μέτρησης και κατά βάση θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος νοοτροπίας μας, ο τρόπος σκέψης μας το μεσαίωνα χρειάστηκε να αλλάξει ο τρόπο σκέψη μα όταν διαπιστώσαμε ότι η γη δεν είναι επίπεδη. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και σήμερα με τον τρόπο που έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα για τα παιδιά ολόκληρου του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much indeed for a very stimulating discussion. Which... Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία είπατε. Ήδη βλέπω κάποια tweet. Το hashtag είπαμε είναι στο 2013. Ωραία. Θα τα δούμε μετά κάποια από αυτά. Τώρα θα ακούσουμε μια ομιλία του Χιμ Στάινερ, το εκτελεστικού διευθυντή του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΟΗΕ και αναπληρωτού Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα μας πει. Ελπίζω να παίξει αυτή τη φορά ο ήχος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι και επιτά μέλη του πάνελ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να μιλήσω στην σημερινή διάλεξη όσον αφορά την βιωσιμότητα της αηφορίας. Όπως φαντάζεστε δεν χρειάστηκε πάρα πολύ προσπάθεια για να πιστώ για τη συμμετοχή μου σε αυτό το πάνελ καθώς θεωρώ πως ο ΙΕ και το πρόγραμμα περιβάλλοντος μπορεί να μοιραστεί κάποια από τα ε, μαθήματα που αντλήσαμε τα τελευταία έτη. Η παγκόσμια αυτή συζήτηση για τη μετάβαση προς μια παγκόσμια οικονομία επηρεάστηκε από την ε, από τις δημοσίευσεις του προγράμματος μας πριν από τρία χρόνια και έκτοτε βεβαίως ε, έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη δημοτικότητα, ηγέτες ε, σε διάφορα υπουργεία, στον ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία των πολιτών έχουν αναγνωρίσει πως πρέπει να υπάρξει μια μετάβαση προς την πράσινη οικονομία, κάτι το οποίο βεβαίω μας οδηγήσει να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε την πρόοδο. Στην Ευρώπη γνωρίζετε τις βασικές τάσεις, θα ήθελα όμως μια στιγμή να εξηγήσω το γιατί η παγκόσμια αυτή συζήτηση είναι τόσο σημαντική και επίκαιρη. Όχι μόνο αντιμετωπίζουμε μία πρόκληση κλιματικής αλλαγής, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης πόρων αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές αλλαγές, κάποιες θεμελιώδεις στο πώς οι οικονομίες μας θα λειτουργήσουν στο μέλλον και όσον αφορά βεβαίως τον αντίκτυπο που έχουν στην δυνατότητα του πλανήτη μας να στηρίξει την ζωή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, σύντομα 10 δισεκατομμύρια, οπότε πρέπει να δούμε τους οικονομικές παραμέτρους αλληλεπίδρασης των οικονομιών, αλλά βεβαίως και την έννοια της αηφόρου ανάπτυξης και κατανάλωσης για να έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος θα μπορέσει να αντέξει ε, πάνω από μία-δύο γενιές. Το έργο του προγράμματός μας είχε στόχο να μπορέσουμε να δούμε μια οικονομική πτυχή των αλλαγών που βλέπουμε τα τελευταία 50 ή και 100 λένε κάποιοι ε, χρόνια. Εξετάζοντας βεβαίως ε, το μέλλον, ε, έχοντας υπόψη ταυτόχρονα την ατμόσφαιρα και την βιόσφαιρα, είναι κατά βάση η βάση της δουλειάς μας. Όμως αυτή τη στιγμή σε υπουργικά συμβούλια, σε κοινοβούλια υπάρχει μία συζήτηση για την ανάλυση κόστους οφέλους. Εδώ πέρα ακριβώς έχει αυξηθεί η ε, περιβαλλοντική διάσταση σε συνδυασμό με μια οικονομική ερμηνεία. Βεβαίως αυτό δεν μειώνει τις επιλογές που έχουμε να κάνουμε. Κάποιες εθικές, κάποιες βεβαίως ε, υπαγορεύονται από τις ε, βασικές οικονομικές οικολογικές με συγχωρείτε, πτυχές της υπόθεσης. Αλλά βεβαίως ε, προσπαθούμε να αποδώσουμε και αξία σε πράγματα τα οποία η φύση μας ε, δίνει δωρεάν θα έλεγε κάποιος ε, παραδοσιακός οικονομολόγος. Η κλιματική αλλαγή και η έκθεση στέρν βεβαίως είναι κάτι το οποίο επιδεικνύει αυτές τις αλλαγές με δραματικό τρόπο. Βεβαίως αυτό θα επηρεάσει και την δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν αλλά και κλάδων ολόκληρων και βιομηχανιών. Αυτή τη στιγμή εδώ στο Ναϊρόμπι συναντάται το Διεθνές Πάνελ για τους Φυσικούς Πόρους υπό την Προεδρία των Ernst Ulrich von Weizsäcker και του Ασοκ Κόσλα. Είναι ένα πάνελ ε, το οποίο υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιληφθούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, όσον αφορά τους φυσικούς πόρους στον πλανήτη τις επόμενες ε, δεκαετίες. Έχουμε λοιπόν δει κάποια πράγματα όσον αφορά το έδαφος, ε, τη χρήση γης, τα μέταλλα. Οπότε η βιώσιμη ανάπτυξη και κατανάλωση, το να αποδώσουμε οικονομική αξία σε κάποια πράγματα, η αποτελεσματική χρήση των πόρων, όλα αυτά ξεκινούν μια συζήτηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Είτε μιλάμε για την Κίνα με την έννοια του οικολογικού πολιτισμού, είτε κάποια νησιωτικά κράτη-μέλη που κινδυνεύουν να χάσουν την επικράτειά τους. Οι ελλείψεις επίσης που αντιμετωπίζει η βιομηχανία ή ζητήματα όπως το νερό, τα μέταλλα, τα ορυκτά και άλλοι βασικοί πόροι της οικονομίας μας. Πώς λοιπόν μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία και πώς μπορεί να μας βοηθήσει η επιστήμη των οικονομικών. Υπάρχουν κάποιες αρχές ε, που είμαι σίγουρος πως και εσείς θα αναφέρετε. Πρώτα απ' όλα τα οικονομικά δεν είναι μια θετική επιστήμη, είναι μια κοινωνική επιστήμη. Οι ε, αγορές λειτουργούν αλλά δεν μπορούμε να πούμε πως υπάρχει κάτι ανάλογο του ε, νόμου της βαρύτητας όταν μιλάμε παραδείγματος χάρη για την προσφορά και τη ζήτηση. Να εξακολουθούμε επίσης να επιδοτούμε την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων με 8 δισεκατομμύρια δολάρια το έτος, ενώ τι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 60 και 70 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αυτό είναι μια επιλογή. Η πρόσβαση στη φτηνή ενέργεια επίσης είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ε, πάρα πολλούς, ενώ για κάποιους άλλους είναι απλά ένα όνειρο. Εδώ όμως στην Κένια, ε, όπου είναι η έδρα του οργανισμού μας, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πράσινης ενέργειας. Είχαμε πάρα πολλές νέες επενδύσεις. 90% των νέων ε, υποδομών αφορά ε, τη γεωθερμική ενέργεια και επίσης ολική ενέργεια και όλο και περισσότερο τα φωτοβολταϊκά. Η υπόθεση λοιπόν αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αντιληφθούμε το πώς οι κυβερνήσεις ε, ως έκφραση της δημοκρατίας μπορούν να αλλάξουν τα μηνύματα στην οικονομία και έτσι η ολόκληρη οικονομία να μετακινηθεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τα οικονομικά της ανανεώσιμης ενέργειας ήδη διαφέρουν πάρα πολύ από ό,τι πριν από 10 χρόνια και έτσι εξηγείται το γιατί στο 2012 υπήρχαν περισσότερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νέες υποδομές, σε σύγκριση με πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα μαζί. Οπότε έτσι μπορεί να γίνει η μετάβαση, αλλά πρέπει βεβαίως να βασιζόμαστε σε επιστημονικά θεμέλια και να έχουμε κατά νου το ρυθμιστικό πλαίσιο, τι τομεακές πολιτικέ και το πώς λειτουργούν οι αγορές. Εάν είναι λοιπόν να μας ακολουθήσει και ο χρηματοπιστωτικός τομέας, πρέπει να δούμε το πώς θα στείλουμε τα σωστά μηνύματα. Θεωρώ λοιπόν πως αυτό είναι το όριο στο οποίο θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, γιατί ο κόσμος έχει λεφτά, αλλά δεν πηγαίνουν αυτά προς την μετάβαση προς την πράσινη οικονομία, αλλά για διάφορους λόγους αποφεύγουν το ρίσκο, τον κίνδυνο. Συχνά ίσως στέλνονται τα λάθος μηνύματα και επενδυτές λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενοι στις πρακτικές του παρελθόντος. Η κλιματική αλλαγή είναι κίνητρο, αλλά ε, δεν μπορούμε να επανεφεύρουμε την παγκόσμια οικονομία μόνο μέσα από το μάτι της βελόνας που είναι η κλιματική αλλαγή. Η επικοινωνία των εθνών και των πραγματικοτήτων στις παγκόσμιες οικονομίες απαιτεί από εμά να διευρύνουμε το ποιες θα είναι οι μεταβάσεις αυτές. Βέβαια, οι προτεραιότητε ενό μικρού νησιωτικού κράτου ή τη Βραζιλία ή τη Κίνα διαφέρουν από αυτέ τη ΗΠΑ ή τη Ιταλία, τη Γερμανία ή τη Δανία. Και μάλιστα, προετοιμάζοντα την έκθεσή μα, βρήκαμε διαφορετικού τρόπου ε, που ακολουθούν διάφορε χώρε προ την πράσινη οικονομία και εδώ πέρα μπορούμε να δεχτούμε από την Ευρώπη ειδικά από το πώ η Ευρώπη βρίσκεται στην πρωτοπορία είτε μιλάμε για την ενέργεια, το μέλλον τη γεωργία, των μεταφορών, των πόλεων, διαχείριση αποβλήτων Όλοι αυτοί είναι τομεί που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να περάσουμε στην πράσινη οικονομία. Ελπίζω με την ΣΤΟΑ να μπορέσετε να συνεχίσετε στην ε, πορεία αυτή για να υπάρξει μεγαλύτερη μετάβαση χωρίς ε, την οποία ο κόσμος θα καταλήξει σε έναν πιο ταλαιπωρημένο πλανήτη και ένα πιο αβέβαιο οικονομικό μέλλον και έτσι ο κίνδυνος μπορεί πλέον να παραλύσει τις επενδύσεις του αντίθετο δηλαδή από αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σε μια εποχή όπου θα πρέπει να έχουμε όχι μόνο ανάπτυξη αλλά και απασχόληση, ποιότητα ζωής κτλ. Και με βάση αυτά θα κριθούμε από τις κοινωνίες. Ελπίζω λοιπόν το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ να συνεχίσει να αποφελείται από την καινοτομία που υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά επίσης να θεωρήσετε και εσείς την δουλειά που κάνουμε στον ΟΗΕ ως κάτι το οποίο μπορεί να αναπτύξει ένα παγκόσμιο, μια παγκόσμια συμφωνία θα έλεγα όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη που μας ενώνει ως μια παγκόσμια κοινότητα κοινωνιών, εθνών και ανθρωπίνων όντων. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στην συζήτησή σας και σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Ε, Έχουμε ένα συμπληρωματικό μήνυμα εδώ. Ε, αν έχετε ερωτήσεις, ε, φυσικά μπορείτε να βρείτε την Διεύθυνση Ελεκτρονικού Ταχυδρομείου και να στείλετε τις ερωτήσεις στον κύριο Στάινερ. Ε, τώρα να πάμε σε μια επόμενη παρουσίαση και πάλι. Μεγάλη ικανοποίηση παρουσιάζω την κυρία Μόνικα Κίρχερ, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος της Infineon Technologies στην Αυστρία και επίσης έχει κάποιες διαφάνειες που θα δούμε σε λίγο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ να παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μια ιδιωτική εταιρεία συγκεκριμένη στο χρηματιστήριο για το πώς εμείς δημιουργούμε θέσεις εργασίας ε, με μια παγκόσμια περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα. Να ξεκινήσουμε με τις κύριες ε, έξι ευρωπαϊκές τεχνολογίες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι υπάρχουν έξι κύριες ε, τεχνολογίες που θα είναι ζωτικές για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τώρα είμαστε ηγέτες ε, σε κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες, αλλά πρέπει πράγματι να τις υποστηρίξουμε και να τις αναπτύξουμε περαιτέρω για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας. Η δική μου εταιρεία δραστηριοποιείται στην ε, μικρο- και νανοηλεκτρονική αλλά επίσης ε, εμπλεκόμαστε ιδιαίτερα στα προηγμένα υλικά και στα προηγμένα μεταποιητικά συστήματα. Γιατί ε, λοιπόν, μιλάμε εδώ για τέτοιες ε, βασικές ε, τεχνολογίες και γιατί εμείς αποτελούμε μέρος αυτού, γιατί βοηθούμε τις υπόλοιπες βιομηχανίες σε σχέση με την παραγωγικότητά τους και την καινοτόμο ισχύ τους. Αν δείτε λοιπόν το κάτω μέρος της πυραμίδας, αυτή τη φορά δεν έχουμε μία πυραμίδα στην Αίγυπτο, αλλά μία αντίστροφη πυραμίδα ή μία αγωγή ευθύνονται για πέντε φορές τον όγκο των πωλήσεων στην ηλεκτρονική και 20 φορές έως 100 φορές σε πωλήσει για την ιατρική ε, βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία κτλ. Ας δούμε τι συμβαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Περίπου 70 ή 80% όλων των καινοτομιών στην αυτοκινητοβιομηχανία έγιναν τις που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες εξαρτώνται απευθείας από την ηλεκτρονική. Αν αυτή η κύρια τεχνολογία λοιπόν δεν υπήρχε πλέον στην Ευρώπη, τότε η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη θα ήταν πολύ χαμηλότερη. Μου λείπει εδώ μια διαφάνεια. Λοιπόν, η ταχύτητα της καινοτομίας ε, τι σημαίνει. Αν ε, το συγκρίνω με το τι συμβαίνει με διάφορους ε, κλάδους, γιατί παίρνει το χάρη ένας αριθμός ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων, ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες και αυτό σημαίνει ότι η δομή τους μικραίνει είναι και περισσότερο η ισχύ ε, των τσίπ διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες. Ε, αν δείτε λοιπόν τι συμβαίνει στο κινητό σας, έχετε την ίδια ισχύ σήμερα που είχε το πρώτο ε, κέντρο ελέγχου της προσελήνωσης. Εάν παραδείγματο χάρη δείτε τι συμβαίνει στις βιομηχανίες των αεροσκαφών, έχει αναπτυχθεί τεράσ... πάρα πολύ το σύστημα αυτό. Ένα Boeing σήμερα θα κόστιζε μόνο 500 δολάρια και θα μπορούσε να κάνει το γύρο του κόσμου μέσα σε 20 λεπτά. Ένα Boeing 767. Βλέπετε λοιπόν ε, ποια είναι η ταχύτητα της καινοτομίας της βιομηχανίας μας. Ε, γιατί χρειαζόμαστε τους ε, ημιαγωγούς στα τσίπ μικροελεκτρονικής για όλες αυτές τις αλλαγές τις επόμενες δεκαετίες. Θα σας φέρω κάποια παραδείγματα, παραδείγματος χάρη ο εξηλεκτρισμός και τα καύσιμα ε, συστημάτων ε, ισχύω. Ε, αυτός ο εξηλεκτρισμός των καυσίμων συστημάτων ισχύω χρειάζεται κάποιους ημιαγωγούς ψηλής ισχύω στα αυτοκίνητα και διπλασιάζεται το περιεχόμενο σιλικόνης ή παραδείγματος χάρη χρειάζεται πολύ μικροελεκτρονική για την ηλιακή ενέργεια για να μπορούμε να έχουμε λειτουργία με έναν οικονομικό τρόπο. Ε, βλέπετε εδώ μία εικόνα από το Facebook, ε, ο μεγάλος αριθμός δεδομένων ε, που έχουμε, όσο μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων έχουμε, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρισμού χρειαζόμαστε. Στη Σιγκαπούρη πριν λίγες ημέρες το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ε, δήλωσε ότι το θέμα της ενέργειας θα είναι ζωτικό ζήτημα ε, και θα δείξει αν η οικονομία μπορεί να τα καταφέρει τις επόμενες δεκαετίες ή όχι. Η Infineon αποφάσισε λοιπόν να επικεντρωθεί σε αυτούς τους τρεις τομείς ενεργειακή αποδοτικότητα, κινητικότητα και ασφάλεια και βλέπουμε μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους για την κινητικότητα, παραδείγματο χάρη, οι αισθητήρε που χρησιμοποιείτε στα αυτοκίνητά σας ε, για την πίεση στα ελαστικά, παραδείγματο χάρη, εγγύονται ένα υψηλό βαθμό ασφάλειας, ε, αλλά και προσωπικής ασφάλειας, ε, γιατί σας ενημερώνουν εγκαίρου αν δεν είναι σωστή η πίεση στα ελαστικά και αποφεύγεται έτσι τα ατυχήματα χρησιμοποιώντας αυτόν τον αισθητήρα. Πρόκειται για ένα προϊόν λοιπόν που αναπτύξαμε και είμαστε σε ηγετική θέση παγκοσμίω ε, με αυτού του αισθητήρε. Έτσι λοιπόν συνδυάζουμε την ασφάλεια και την προσωπική ασφάλεια αλλά και την κινητικότητα ή για τα κινητά σα ή για τα λάπτοπ παραδείγματο χάρη. Ε, υπάρχει ένας ε, μηχανισμός ε, ταυτοποίησης που θα είναι όλο ένα και πιο σημαντικό σε σχέση με την ασφάλεια. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ελεπίδραση μεταξύ αυτών των τριών τομέων εστίασης, αλλά θα επικεντρωθούμε σήμερα περισσότερο στην ενεργειακή αποδοτικότητα. γιατί με αυτό το θέμα ασχολούμαστε κυρίως, με αυτό το τομέα ασχολούμαστε κυρίως στην Ινφίνων Αυστρία. Έχουμε λοιπόν χαράξει τη δική μας στρατηγική και αποφασίσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με έναν αηφόρο τρόπο για τις επόμενες δεκαετίες. Χρειαζόμαστε αυτούς τους πέντε τομείς ανταγωνιστικότητας να βρίσκονται στο επίκεντρό μας συνέργεια και αυτή καθ' αυτή, ηγετική θέση στην κοινοτομία, βρίσκεται στο κέντρο. Επίσης μας ενδιαφέρει η αριστεία των εργαζομένων και επίσης και οι ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης που έχουμε ε, και βλέπετε δεξιά και αριστερά έχουμε την αριστεία στην ποιότητα και στο επιχειρηματικό σκέλος και έχουμε ε, και ανάλογες και μικτές ε, αρμοδιότητες. Έχουμε ένα παράδειγμα για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα σας δώσω αργότερα τις διαφάνειες. Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Πράσινη βιβλία για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τότε εμείς εκπονήσαμε κάποια παραδείγματα για το πώς η μικροελεκτρονική θα μπορούσε να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα σε διάφορες εφαρμογές. Και ανακαλύψαμε ότι παραδείγματο χάρη για ε, την ηλεκτρική ενέργεια γενικά μέχρι και υπήρχε δυναμική εξοικονόμηση μέχρι και 34%. Αυτό μπορούσαμε να το πετύχουμε χρησιμοποιώντας ε, τα τελευταία τεχνολογία. Έτσι λοιπόν, ε, χάνεται 34% ενέργεια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επειδή δεν χρησιμοποιούνται οι τελευταίες τεχνολογίες για το φωτισμό. Ε, φτάνουμε από το 20 μέχρι το 30% της ενέργειας που χάνεται τώρα γιατί δεν χρησιμοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογίες και μπορώ να συνεχίσω έχουμε το χάρη και τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις τηλεοράσεις και άλλες εφαρμογές. Έτσι λοιπόν ε, το δικό μας προϊόν μπόρεσε να αυξήσει τα επίπεδα ζωής σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας αλλά βλέπετε εδώ και κάποια αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την εταιρεία μας. Χρησιμοποιούμε 34% λιγότερο νερό για να παρασκευάσουμε ένα ε, εκατοστό δίσκου ημιαγωγού από ότι ο παγκόσμιο μέσος όρος και καταναλώνουμε 44% λιγότερες ενέργειες για τον ίδιο δίσκο ημιαγωγού. Έτσι λοιπόν εμείς ε, υποστηριζόμαστε και από ένα ε, ουδέτερο ερευνητικό κέντρο και αυτό σημαίνει ότι δίνουμε πάρα πολλά προϊόντα στη βιομηχανία παγκοσμίω και καταλήγουμε στο εξής. Ε, τελικά έχουμε λιγότερους ε, τόνους διεξιδίου του Αφρικά 15,8 εκπο... τόνους σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα λιγότερους. Τώρα υπάρχει και ένα σημαντικό θέμα που δεν πρέπει να υποτιμάμε. Μεγάλες ε, εταιρείες ε, στην Ευρώπη εργάζονται κατά μήκος της ελισίδας ε, αξίας. Έτσι λοιπόν, αυτά τα 560 εκατομμύρια ευρώ του όγκου αγορών πέρσι επενδύθηκαν σε συμπράξεις, σε πολλές μικρές και μεσές επιχειρήσεις ε, στην περιοχή. Ε, έτσι λοιπόν ε, πολλές ε, φορές ε, μικρές και μεγάλες εταιρείες μαζί με πενεπιστήμια συνεργάζονται για να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή και αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Ρούμπικ ήταν ότι θα ήταν καλή ιδέα να κάνουμε μια έρευνα για το θέμα αυτό γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε περισσότερο τι γίνεται στις αλυσίδες αξίας σε όλα τα στάδια και με όλες τις εταιρείες που συνεργάζονται. Τώρα έχουμε ηγετική θέση στον τομέα της ε, καινοτομίας. Αυτό σημαίνει όχι μόνο να προβαίνουμε σε έρευνα και σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά εδώ και 7 χρόνια έχουμε υιοθετήσει ένα καλό σύστημα καινοτομίας ε, και έχουμε δημιουργήσει μια συγκεκριμένη κουλτούρα Θέλω να επικεντρωθώ στην ε, ενεργή διοίκηση, μεταφορό, διαχείριση μεταφοράς. Τι σημαίνει αυτό, ότι τελικά υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρουμε νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα σε άλλες εταιρείες, σε άλλους εταίρους, σε άλλες τοποθεσίες και να δημιουργήσουμε χώρο για νέα οργανωτική αλλά και κοινωνική καινοτομία. και να πω τα αποτελέσματα ήταν 400 mm ισχύω που είχαμε. Τα, ε, το εργατικό δυναμικό με το ταλέντο του μπορεί να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις και να δει ποιε είναι οι νέε δυνατότητε στην αγορά εργασία. Επομένω, προσλαμβάνουμε ανθρώπου από όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε εργαζομένους που προέρχονται από 55 χώρες και στην ε, Καρινθία είμαστε σε ηγετική θέση σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των τεχνικών. και χρησιμοποιούμε ερευνητέ ε, με πολύ υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχει ιδρυθεί και, ένα και μια διεθνής ε, σχολή προκειμένου να ε, μπορούμε να εφαρμόζουμε τις προσεγγίσεις της καινοτομία μας και εκεί πέρα από το τεχνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. No, I think the technical problems are more on ε, μάλλον εμείς πρέπει να σας ζητήσουμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα. Ίσως χειρίσουμε σε πιο παραδοσιακές μεθόδους. Δηλαδή να αρχίσουμε να ζητάμε από κάποιον ε, την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, όπως κάναμε παλιά. Μας περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ Μονικά. Θα ήθελα πριν περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση να σας ενημερώσω ότι είχαμε ήδη λάβει κάποιες ερωτήσεις. Ευχαρίστως να δεχτούμε κι άλλες και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αμέσως μετά. Εάν δεν είχατε πάρει προμηθευτεί αυτό το χαρτί για την υποβολή ερωτήσεων, σας προτείνω να το πράξετε και να το ε, σηκώσετε το χέρι σας έτσι ώστε κάποιος να το φέρει εδώ στο Προεδρείο. Και να αποβάλλετε έτσι την ερώτησή σας. Προχωρούμε λοιπόν στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Hans Πράνιξ, εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Έχετε το λόγο, Hans. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω τα τεχνολογικά εργαλεία. Αν δεν ε, δουλέψει θα ζητώ και εγώ να προχωρούμε στην επόμενη διαφάνεια από τον τεχνικό μας. Μπορώ να βλέπω τις διαφάνειες στην οθόνη μου, ρωτάει ο μιλητής. Ωραία. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Επομένω είναι μάλλον προφανές ότι εμείς εστιαζόμαστε στο ε, επίθετο πράσινη όταν μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη. Αναφερόμαστε δηλαδή στο περιβαλλοντικό, στην περιβαλλοντική πτυχή της πράσινης ανάπτυξης και όπως σε πολλές άλλες πολιτικές θα έπρεπε να θέσουμε στόχους όλο και πιο φιλόδοξους. Ας εξετάσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο καταρτίζεται η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική πολιτική μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν τρία στάδια χρονικά. Πρώτα απ' όλα αυτό που κάνουμε καθημερινά, δηλαδή να επιδιώκουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο στα περιβολικά δεδομένα, δηλαδή όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του ύδατος, του νερού κτλ. Ε, για τα στοιχεία για τα οποία υπάρχουν ήδη κανονισμοί και οδηγίες. Όπως όμως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια φιλόδοξη στρατηγική έως το 2020, η οποία συνεχίζεται για το 2030 και έχουμε ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους μέχρι το 2050. Άρα μιλάμε ήδη για στόχους μέσω μακροπρόθεσμος, Πέρα από την καθημερινή και βράχη πρόθεσμη παρακολούθηση. Για εμά ε, στην υπηρεσία είναι εξαιρετικά σημαντικό η δημιουργία η κατάρτιση τη στρατηγική για το 2050, η οποία προσπαθεί να αντικατοπτρίσει τρει κυρίε ιδέε. Πρώτα απ' όλα τη συμμετοχή τη τοπική κοινωνία, δεύτερον την κυκλική οικονομία ε, χαμηλών, χαμηλής αξιοποίησης ε, των φυσικών πόρων και τρίτον την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων. που είναι και ένα ξεχωριστό ζήτημα, η ε, ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων δηλαδή. Κοιτώντα τις επιδιώξεις μας το 2050, θεωρούμε ότι δεν αρκεί ο τρόπος σκέψης που ακολουθούσαμε και μέχρι τώρα και οι πολιτικές που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα, οι οποίες βασίζονταν μόνο στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. Επομένως είναι μεταβατική αυτή η εστίαση στην αποτελεσματικότητα. Τρία είναι τα κύρια στοιχεία που έχουμε στο μυαλό μα σε σχέση με την πράσινη οικονομία. Η χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, η κυκλικότητα της οικονομίας ε, που κάνει μικρή χρήση των φυσικών πόρων και τρίτον αυτό που σας είπα για την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων. Στη διαφάνεια αυτή, στη γράφημα αυτό, ε, σας ε, παρουσιάζω το Human Development Index, το δίκτυο ανθρώπινης ανάπτυξης. Εάν αυτός είναι πάνω του 0,8% μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά κάποιο απολαμβάνει τη ζωή του. Η πρόκληση λοιπόν που αντιμετωπίζουμε είναι ότι η παραδοσιακή προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ποιότητα ζωής πλέον αρχικά πηγαίνοντα και αξιοποιώντα και καταχρώντας μάλλον τους, ε, καταχρώμενοι τους φυσικούς πόρους και μετά αφού επιτύχουμε αυτή την ευζοία με έναν μαγικό τρόπο να εφαρμόσουμε πολιτικές αηφορίας και ξαφνικά να πέσουμε σε χαμηλή ε, κατανάλωση και χρήση των φυσικών πόρων. Όμως, αν κοιτάξουμε το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν ήμασταν επιτυχείς. Αυτός ο τρόπος, αυτή η μέθοδος δεν ήταν επιτυχής. Άρα πρέπει να βρούμε μια άλλη. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Δεύτερο, δεύτερη απάντηση που δίνω στο ερώτημα γιατί πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά τώρα. Μπορούμε να ε, πάμε μια διαφάνεια πριν παρακαλώ. Εάν γίνεται αυτό, ρωτάει ο μιλητή. διάλεξε στόα. Είναι φαντάζομαι τα τεχνολογικά εργαλεία θα έπρεπε να λειτουργούν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ω περιβαλλοντική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώ ε, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα το πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον. Το οποίο στον τίτλο του αναφέρεται στα οικολογικά όρια. Επομένω, ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δουλειά μα βασίζεται σε τρεις ομόκεντρους κύκλους, ομόκεντρους κύκλους που καθορίζουν τα όρια, δηλαδή τα οικοσυστήματα, τα κοινωνικοτεχνολογικά συστήματα. Εμείς εστιάζουμε, μάλλον, θεωρούμε ότι τα οικοσυστήματα θέτουν τα όρια από την περιβαλλοντική πλευρά και τα κοινωνικοτεχνικά συστήματα καθορίζουν ποιες είναι οι οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, τις οποίες δεν διαχωρίζουμε μεταξύ τους λαμβάνουμε όψη μας όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπετε εκεί, την πολιτική, τις αξίες, την τεχνολογία, την επιστήμη, την ανάγκη της αγοράς, τους κλάδου της βιομηχανίας, γιατί προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία ε, αλληλεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους. σε παγκόσμιο επίπεδο αναφέρθηκε πριν και ο κ. να έχουμε τους, τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Τον Ιούλιο είχαμε την ε, αξιολόγηση που μας έδειξε ότι όσον αφορά τους οικονομικούς στόχους ε, έχουμε βρεθεί σε αρκετά καλό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει μείωση της φτώχειας, για παράδειγμα, πολέμηση της φτώχειας. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στους περιβαλλοντικούς στόχους, στην περιβαλλοντική πτυχή των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Τι λείπει όμως εδώ, η σχέση αιτίου αιτιατού. Δηλαδή καταφέρνουμε να μειώσουμε, να καταπολεμούμε την φτώχεια με τρόπο μη αηφόρο, με τρόπο που βλάπτει το περιβάλλον. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση μεταξύ αυτών των δύο ομάδων στόχων και γι' αυτό χρειάζεται να δούμε το ζήτημα του περιβάλλοντος και τη σχέση τους με τις πολιτικές μας πιο θεμελιωδώς, πιο ε, εις βάθος. Εδώ βλέπουμε την αγοραστική δύναμη, η οποία προφανώς σχετίζεται με την προσφορά και τη ζήτηση. Βλέπουμε ότι αυξήθηκε κατά 2,5 φορές. Η μεσαία τάξη αυξάνεται ραγδαία, ιδιαίτερα στην Ασία και τον Ειρηνικό ωκεανό, σε αυτή την περιοχή. Και μας εκπλήσει το γεγονό ότι ξαφνικά θεωρούμε πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίες δεκαετίες αυτή τη μεσαία τάξη. Ε, ενώ ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να καταφέρουν μέσω της εκπαίδευσης, μέσω των ευκαιριών, μέσω των ευκαιριών επασχόλησης που θα είχαν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Εδώ που τα λέμε, εκεί θα έπρεπε να στοχεύουμε ως άνθρωποι. Δηλαδή έναν τρόπο ζωής που να προσυδειάζει με αυτόν της μεσαίας Δεδομένα, λοιπόν, δεδομένων λοιπόν όλων αυτών των στοιχείων, η στρατηγική για το 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας οδηγεί πράγματι σε μια πράσινη οικονομία. Γιατί θέτει μια σειρά στόχων για την βιοπικιλότητα, για το περιβάλλον, για την ποιότητα του αέρα και του νερού, καθώς επίσης και διάφορες πρωτοβουλίες για την πράσινη οικονομία, εγκάρσεις πρωτοβουλίες, που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε λοιπόν λοιπόν να σκεφτούμε το επόμενο βήμα, πώς ε, αυτή η στρατηγική μέχρι το 2020 θα μετεξελιχθεί σε μια στρατηγική μέχρι το 2030. Ε, θεωρούμε ότι μέχρι τώρα αυτή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή, αυτό το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στιαζόταν στην αποτελεσματικότητα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, την κατανάλωση ενέργειας. Τέσσερις διαφάνειες έχω ετοιμάσει για την κατανάλωση ενέργειας. Ε, η σε αυτά τα γραφήματα αυτά η πάνω πάνω γραμμή, η καμπύλη είναι πάντα η οικονομική αποτελεσματικότητα και η κάτω κάτω γραμμή είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ε, η μεσαία γραμμή είναι συνήθως οι πρώτες ύλες που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν. Αναφέρομαι κυρίως στην Ευρώπη. Εδώ η αποσύνδεση των δύο στοιχείων είναι κάπως μεσαίου ε, επίπεδου στην Ευρώπη. Στο μέλλον, εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε τέτοιες πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή η αποσύνδεση θα πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερη. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, αλλά παραμένουν τα όρια όσον αφορά τους φυσικούς πόρους. Εδώ σα φέρω ένα παράδειγμα σε σχέση με την αυτοκίνητο βιομηχανία με τα οχήματα. Ε, αυξάνεται η χρήση του αυτοκινήτου όπω αυτή αντικατοπτρίζεται από το συνολικό αριθμό χιλιόμετρων που ε, διανύονται με, με, με αυτοκίνητα. Μειώνεται η κατανάλωση ε, καυσίμων, καλό αυτό. Μάλλον, με συγχωρείτε, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα, αλλά αν δούμε συνολικά την κατανάλωση καυσίμων, αυτή αυξάνει. Γιατί αυξάνεται και ο αριθμό του. Με άλλα λόγια, όσον αφορά τις μεταφορές, δεν αρκεί η αποτελεσματικότητα. Μπορεί να μου πείτε ότι ναι, αυτό απλώς θα αλλάξει όταν θα έχουμε τη τεχνολογία στη διάθεσή μας που θα μας δώσει τη δυνατότητα όλοι να χρησιμοποιούμε υφρυτικά. Αν όμως όλοι χρησιμοποιούμε. Εάν όλοι λοιπόν φτάσουμε να χρησιμοποιούμε 100% ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα παραμείνει το πρόβλημα ε, αν αυξάνεται ο αριθμό των αυτοκινήτων. Θα παραμείνει το, πρόβλημα ε, στις, στι ίδιε ίδιες τις μεταφορές, τα ποντιλιαρίσματα. Σε μια πράσινη οικονομία το ιδιωτική χρήση αυτοκίνητο θα παραμείνει να έχει έναν σημαντικό ρόλο, αλλά θα έχει αλλάξει αυτό ο ρόλο. Βλέπετε εδώ μια φωτογραφία από ένα μποτιλιάρισμα στην ε, Οδόντε Λαλουά την, την μεγαλύτερη οδική αρτηρία των Βρυξελών. Μακάρι να μην έχουμε μια τέτοια εικόνα στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν αστιάσει στην αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων. Και έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, την οποία σημειώνουμε το πράσινο κίτρινο ε, σημειώνει την ε, μέτρια πρόοδο και το κόκκινο είναι τα θέματα στα οποία έχουμε ακόμα πρόβλημα. Εάν εξετάσουμε την μείωση των εκπομπών ε, των αερίων που προκαλούν φαινόμενο του είμαστε καλά. Αλλά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των οικοσυστημάτων, την ανθεκτικότητα μάλλον των οικοσυστημάτων, κατά πόσον αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ε, προκλήσεις που του θέτει η χρήση αυτών των οικοσυστημάτων από την κοινωνία, βλέπουμε ότι εδώ είμαστε στο κόκκινο. Η πρόκληση λοιπόν είναι να μην συνεχίσουμε να εστιάζουμε τόσο πολύ στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. με αυτή η αύξηση της αποτελεσματικότητας είναι σημαντική, αλλά ουσιαστικά πρέπει να επιδιώξουμε μια συστημική αλλαγή, μια συστημική βελτίωση προκειμένου να μεταβούμε προς την πράσινη οικονομία. Αυτό έχει επιπτώσεις και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι επενδύσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις δηλαδή, και στον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα, ένα εκατομμύριο δολάρια. Μπορούμε αυτά να τα επενδύσουμε είτε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, δηλαδή για παράδειγμα για ένα ιδιωτική χρήση αυτοκίνητο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της μηχανής εσωτερικής καύσεως του ή να τα επενδύσουμε σε κάτι που θα είναι τελείως, διαφορετικό, τελείως καινοτόμο και το οποίο θα μας βελτιώσει το σύστημα συνολικά. Επομένως, επιδιώκοντας τους στόχους μέχρι το 2020 δεν πρέπει να ε, δημιουργήσουμε για τους μας αδιέξοδα τα οποία θα μας αποτρέψουν από το να πετύχουμε τους στόχους μας για το 2050. Θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το 2020 με την αποτελεσματικότητα, αλλά αν όλες οι επενδύσεις πάνε προς την αποτελεσματικότητα, πώς θα καταφέρουμε μετά έως το 2050 να επιτύχουμε τους στόχους που θέτουμε για το 50 που θα είναι τελείως διαφορετική, που θα είναι πλέον για, μιλούν πλέον για μείωση των ορυκτών καυσίμων συνολικά. Επομένω πρέπει να σκεφτούμε την μετάβαση θεμελιώδεις αλλαγές όχι μόνο στο τεχνολογικό πεδίο αλλά επίσης στον τρόπο ζωής, στις δομές, της κοινωνίας και ε, οτιδήποτε, οποιαδήποτε επίπτωση έχει αυτό στην καθημερινότητά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προετοιμάσει έναν οδικό χάρτη έως το 2050, μια σειρά μάλλον οδικών χαρτών έως το 2050 που αναφέρονται στην ανταγωνιστική οικονομία χαμηλού εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρακα το 2050, μια, ένα οδικό χάρτη για την ενία ε, χώρα μεταφορών, έναν οδικό χάρτη για την Ευρώπη με αποτελεσματική χρήση των πόρων και έναν οδικό χάρτη για την ενέργεια ως το 2050. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που έχουμε. Στη διαφάνεια αυτή διαπιστώνουμε ότι αρχίζει να υπάρχει ένα πρόβλημα που θα πρέπει να το ε, επιλύσουμε για να καταφέρουμε μέχρι το 2050 να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας. Με την κόκκινη γραμμή βλέπετε που μας οδηγεί η τρέχουσα πολιτική. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα επιτύχουμε αποτελεσματικότητα συνολικά σε όλο τον κύκλο της παραγωγής. Ε, ε τώρα έχουμε εστιάσει στην αποτελεσματικότητα στην, στην κατασκευή, στη χρήση των φυσικών πόρων, στη χρήση των πρώτων υλών. Όμως πρέπει να ασχοληθούμε τώρα και με ζητήματα για παράδειγμα την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων. για να αντιμετωπίσει η κοινωνία τις μελλοντικές προκλήσεις. Με ποιον τρόπο λοιπόν μπορούμε να καταρτήσουμε πολιτικές που θα υποστηρίζουν αυτή τη μετάβαση. Θα πρέπει να σταματήσουν να υφίστανται οι επιδοτήσεις οι οποίες βλάπτουν το περιβάλλον. Αναφέρθηκε ήδη η επιδότηση παραδοσιακών καυσίμων. Η τελευταία έκθεση του ΑΣΕ αναφέρεται σε 1,3 ε, εκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν και θα έπρεπε να αξιοποιούνται αλλιώ. Θα πρέπει αντιθέτως να αναπτύξουμε για να ενθαρρύνουμε όχι μόνο τεχνολογίες αλλά και πρακτικές οι οποίες ε, πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της πρακτικής οικονομίας και σημαντικό στοιχείο σε αυτό είναι η ε, ανταλλαγή γνώσης που αναφέρεται σε, αυτές, σε αυτή τη μετάβαση έχουμε ένα πενταετές πολυετές σχέδιο με το οποίο θα ασχοληθούμε για παράδειγμα στο ζήτημα της ποιότητας ζωής με τη σχέση μεταξύ υγείας, κατανάλωσης και χημικών. Ε, υπάρχει το ζήτημα των δικτών που ήδη αναφέρθηκε. Ε, προσπαθούμε να ε, συμπεριλάβουμε οικολογικούς δείκτες στον τρόπο με τον οποίο η Eurostat μετρά ε, τα, τα στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη και προφανώς συνεργαζόμαστε και με το πρόγραμμα το περιβαλλοντικό του ΟΗΕ. Μια πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πώς θα συνδέσουμε αυτές τις στρατηγικές έως το 20 και έως το 30 με τη γενικότερη στρατηγική μας μέχρι το 2050. Για να μπορέσουμε το 2050 τελικά να επιτύχουμε αυτό που θα θέλαμε. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί μετάβαση θεμελιώδη σε όλα τα κοινωνικά και τεχνολογικά επίπεδα. Αυτό επίσης σημαίνει ότι θα χρειαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο πιο αποτελεσματική δράση. Η Ευρώπη δεν είναι απομονωμένη, αλληλεπιδρά με τον υπόλοιπο κόσμο, ιδιαίτερα οικονομικά αλλά και αλλιώς. Θα πρέπει μάλλον να υπάρξει μια πολύ θεμελιώδης αλλαγή όσον αφορά το μήνυμα που διατυπώνουμε, το λόγο που διατυπώνει η Ευρώπη. Αναφέρθηκε και σήμερα ένα παράδειγμα. Είπαμε ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις επόμενες γενναίες όταν ε, σκεπτόμαστε και καταπτύσσουμε αυτές τις πολιτικές. Αλλά εγώ έχω μια ένσταση όσον αφορά αυτές, αυτή την ορολογία. Ε, όταν αναφερόμαστε στις επόμενες γενναίες στον πληθυντικό είναι σαν να νομίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε ακόμα μια γενιά μέχρι να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα. Ε, δεν ισχύει αυτό. Αν μιλάμε για τη στρατηγική για το 2050 καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να καταφέρουμε να ζήσουμε το μισό της ζωής μας, το μισό της ζωής ενός παιδιού σήμερα ε, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο θα έχει ε, ε, ανθεκτικά οικονολογικά συστήματα και μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης φυσικών πόρων. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει σήμερα, ήδη από τώρα και αυτό ήταν νομίζω το κύριο μήνυμα που θα ήθελα να σας δώσω. Ευχαριστώ. Well, thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές μας. Έχουμε μισή ώρα τώρα για ερωτήσεις. και η πιο σημαντική ανακοίνωση σήμερα είναι πως μετά θα σερβίρουμε ποτά. Οπότε έτσι μπορεί να μην ακούσουμε πολλές ερωτήσεις αναλόγως. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις ήδη, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από τον Χωσέ Φανάνισελ Χόβεν, την Χωσέ, με συγχωρείτε, πρώην Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ράντναρ, να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Θυμάστε ποια ήταν η ερώτηση που θέλατε να κάνετε. Ναι, λοιπόν, να ρωτήσω τον κύριο Ισμαήλ Σεραγγελτίν. Θεωρείτε πως ο ανθρώπινος παράγοντας έχει τύχει αρκετής προσοχής στις ομιλίες των άλλων ομιλητών. Ή μήπως αλλάζουμε ήδη την οπτική μας προς την κατεύθυνση που θεωρείτε εσείς σωστή για το μέλλον. Και η συνάδελφος βεβαίως θα συνοψίσει στο τέλος, αλλά μπορεί να απαντήσει. Σύντομα, ναι. Θεωρώ πως αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και νομίζω πως μόλις βλέπουμε πως γίνεται κάποια δουλειά με τη Eurostat και τα λοιπά, γιατί θεωρώ πως εάν είναι ε, λάθος τα μηνύματα, λάθος θα είναι και οι πολιτικές. Ανεξαρτήτως του ποιος είσαι. Γι' αυτό χρειάζονται καλύτερα στατιστικά στοιχεία. Η ανθρώπινη πτυχή δεν αναφέρθηκε αρκετά. Αλλά υποθέτω πως θα ληφθεί υπόψη. Θα σας πω όμως πως είχαμε πολλές δυσκολίες στο να βρούμε παρκείς ορισμούς του κοινωνικού κεφαλαίου. Εγώ, ο Ντασγκούπτα και πάρα πολλοί άλλοι ε, ασχοληθήκαμε με αυτά τα ζητήματα, αλλά τώρα όλοι αποδέχονται την ανθρώπινη πτυχή. Παρακολουθείτε με πολλούς τρόπους Υπάρχουν γραφήματα που δείχνουν την ποιότητα της υγείας, ε, της εκπαίδευσης, που είναι εξίσου σημαντική με την ποσότητα. Βασικό παράδειγμα, η που ξοδεύει πολύ περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον στην υγεία, ξοδεύουν, και έχουν πιθανότατα τα χειρότερα αποτελέσματα σε, από τις προηγουμένες χώρες. Η πρώτη σημασία έχει και το αποτέλεσμα και πώς το επιτυγχάνουμε. Και πολλή δουλειά γίνεται εκεί πέρα. Σημασία λοιπόν έχει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να πάμε προς τα εκεί. Σας ευχαριστώ. Να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις ακόμα. Θα δώσουμε ευκαιρία σε όλα τα μέλη να μιλήσουν. Ας ακούσουμε τώρα τον κύριο Λάμπρεχτς. Εδώ είναι? Ναι. Θέλετε να κάνετε την ερώτησή σας. Ναι, στο πρώτο βίντεο οι ευρωβουλευτές μίλησαν για το ότι θα πρέπει αυτοί που χαράσουν την πολιτική να διαμορφώνουν προδιαγραφές και οι, ε, αυτοί που καινοτομούν να καινοτομήσουν. Η ερώτησή σας, η ερώτησή μου ποιος είναι ο ρόλος ε, αυτών που καινοτομούν στην Αυστρία, στην Ευρώπη και στις συζητήσεις που γίνονται τώρα στη Βαρσοβία. Ο ρόλος αυτών που χαράζουν πολιτική είναι πρώτα να έχουν ένα όραμα για την Ευρώπη και μετά να γίνει αυτό μια στρατηγική. Η στρατηγική η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει βεβαίως τους ε, βασικού ενδιαφερόμενους, όχι μια στρατηγική ε, ερήμην ε, του τεχνολογικά εφικτού και βεβαίως το, αυτό που με απασχολεί πολύ το εκπαιδευτικό σύστημα γιατί στατική και όραμα θα υλοποιηθούν μόνο αν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν. Υπήρχε και ένας νομπελίστας που είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τα πάντα σωστά αλλά πάρα πολύ αργά. Οπότε, αν είναι να μιλάμε για μια μελλοντική στρατηγική πρέπει ταυτόχρονα να ε, υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα την εφαρμόσουν τη στιγμή που τη γράφουμε. Κάποιος άλλος θα ήθελε να σχολιάσει. Όχι, ωραία. Έχω εγώ μια ερώτηση προς τον Hans Μπράνινγκς από τον Κόεν Ελσαμάν. Κάνετε την ερώτησή σας. Ναι. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, για την ομιλία σας. Πολύ ενδιαφέρουσα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν γιατί είστε τόσο αισιόδοξο για το 2050. Όταν βλέπουμε μετά στις διαφάνειες ένα τεράστιο κενό μεταξύ των ε, τωρινών πολιτικών και των τελικών στόχων μείωσης των εκπομπών. Οπότε ε, θετικό το μήνυμά σας, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει στο πλαίσιο της οικονομίας και της πολιτικής για να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί. Γιατί είμαι αισιόδοξο. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι αισιόδοξο. Είναι ηθικό καθήκον όπως συχνά λέγεται. Και τη δική σας γενιά νομίζω πως είναι καθήκον της γενιάς μου να είναι αισιόδοξη, αλλά επίσης είμαι αισιόδοξο για πολλούς άλλους λόγους. Πρώτα απ' όλα, αν ακούσετε τη συζήτηση τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρώπη, όπου πολλοί λένε πως από την κρίση του 2008 δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για για νέες πρωτοβουλίες και πιεζόμαστε η ανάπτυξη για δουλειές. Μα τα τελευταία πέντε χρόνια προέκυψε η ατζέντα για το 2050. Ακόμα λοιπόν και αν υπάρχει ένα οικονομικό ζήτημα που δεν το αγνοώ, το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα προχωράει και τα καταφέρνουμε στην Ευρώπη και σε παγκόσμια κλίμακα να καθορίσουμε τη συζήτηση. Αυτός είναι ένας λόγος αισιοδοξίας δεύτερον. Έχουμε τώρα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το 2050 που είναι ένα πρόγραμμα μετάβασης πριν από 10 χρόνια. Ως επιστήμονες έπρεπε να φέρουμε αυτή την οτροπία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μας έλεγαν αυτά είναι επιστημονικά, τραβηγμένα ή μη ρεαλιστικά κτλ. Τώρα έχουμε έγγραφα πολιτικής τα οποία μπορούμε να αναφερθούμε. Οπότε, εάν μπει αυτό στο πενταετές πρόγραμμα εργασίας μας, δεν μπορούν να πούνε στις Βρυξέλλες «Μα τι κάνουν αυτοί στην Κοπενχάγη». Όχι, απαντάμε σε αυτά τα οποία μας λέτε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πολιτικό ε, βήμα αυτό το οποίο έχει γίνει. Ένα τρίτο στοιχείο είναι πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν πως το θέμα δεν είναι να είμαστε μη ε, Το μη ρεαλιστικό είναι να συνεχίσουμε με την ε, τωρινή, το τωρινό σύστημα κατανάλωσης και παραγωγής, ε, το οποίο δεν είναι πλέον αηφόρο. Και κάτι τέτοιο είναι ανέθυνο. Αν δεν αλλάξουμε κατεύθυνση, ε, θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση μη βιώσιμη. Οπότε είναι σαφές πως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πράγματα εκ βάθρων. Και αυτό φαίνεται και στα έγγραφα πολιτικής. Αν δούμε τώρα την οικονομία. Νομίζω πως ε, υπάρχουν ε, εταιρείες, ε, φορείς, καινοτόμοι άνθρωποι που σκέφτονται με τρόπο πρωτότυπο και βασίζονται σε μια νέα νοοτροπία και είναι επιτυχής. Εκεί πέρα λοιπόν αναζητώ αισιοδοξία και ο άλλος λόγος αισιοδοξία. Και αυτό δεν το λέω γιατί είστε νέο. Μέχρι πριν από πέντε μήνε πριν αναλάβω αυτή τη δουλειά, ήμουν καθηγητής και κάθε χρόνο έκανα ένα μάθημα για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Όταν έχετε κανείς σε επαφή με τους νέους ε, και βλέπει αυτές τις ιδέες από το αμφιθέατρο και ο κόσμος σκέφτεται το μέλλον του, ε, είμαι αισιόδοξο. Αλλά, αλλά και ρεαλιστή. Έχουμε πολλή δουλειά και είναι διαρθρωτική δουλειά που πρέπει να γίνει. Δεν είναι στα περιθώρια. Δεν είναι μόνο θέμα αύξησης αποτελεσματικότητα. Θεωρώ λοιπόν πως τώρα μπορώ να συνεισφέρω τουλάχιστον ε, στη... στο να επηρεάσω την πολιτική και την σκέψη. Σας ευχαριστώ. Τώρα, στο Twitter γίνεται χαμός, κυρίως από κάποιους. Και θα ήθελα να ακούσουμε τώρα μία ερώτηση από τον Σάιμον Σεφ από το Πανεπιστήμιο του Ψάλα. Είναι εδώ? Α, εσείς είστε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την αισιοδοξία. Αυτό χρειαζόμαστε. Κοιτάζοντας το έγγραφο Τη διάσκεψης του Ρίο Συν 20 πέρσι βλέπουμε καλές προθέσεις αλλά και ανοιχτούς ορισμούς για το τι είναι η πράσινη οικονομία και η μετάβαση προς αυτήν. Και νομίζω πως λογικό είναι να μιλάμε για μια μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί τα προβλήματα είναι παγκόσμια. Και μετά, να δούμε τις αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία, οι χώρες αυτές έχουν ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 10%, πάνω από το 10% που δεν μπορούν να διατηρηθούν. Και πώς νομίζετε, πόσο, ρε, πόσο ρεαλιστική νομίζετε πως είναι η μετάβαση σε μια παγκόσμια πράσινη οικονομία με βάση αυτά και πώς μπορεί να το επηρεάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. James Lozzi επίσης, ο οποίος ε, είναι στο Twitter και έχει κάνει κάποιες παρόμοιες ερωτήσεις. Πώς μπορεί να τα επηρεάσει αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τα μέλη του πάνελ μας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια σταδιακή επιβράδυνση ε, αυτών των μεγεθών ανάπτυξη. Όμω το σημαντικό είναι πώ μετρώνται, χωρί να λαμβάνονται υπόψη, παραδείγματο χάρη, το υψηλό κόστο τη ρήπανση ε, στην Κίνα και είδαμε ποια είναι τα ποσοστά ανάπτυξης στην Ινδία από το συνάδελφο και ότι αυτά δεν ε, βρίσκουν αντίκτυπο στη ζωή πολλών ανθρώπων. Όμως, αν δούμε τι συμβαίνει σε ορισμένες πλούσιες χώρες σε σύγκριση με κάποιες αναδυόμενες αγορές ή αναπτυσσόμενες χώρες, το ποσοστό των πόρων που χρησιμοποιούνται αναμονάδα του ΕΚΠΕ ή των εκπομπών ανα μονάδα του ΕΚΠΕ είναι πολύ πιο μειωμένο στις προηγμένες χώρες εν μέρη. Αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί να έχουμε με τόσο χάρη 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα και, και άνθρακα ή ξύλα για να ζεσταθούν, αλλά αναμονάδα του ΕΚΠΕ βλέπουμε μείωση συν χρόνο. Τώρα, αν ε, πράγματι Είμαστε επιτυχεί στην επόμενη μετάβαση, στην οποία αναφέρθηκε ο Χάνς, ε, που θα έχει να κάνει όχι με την αποδοτικότητα, αλλά με την μεταμόρφωση των ε, οικοσυστημάτων. Τότε, όχι μόνο θα έχουμε μία καλύτερη δυνατότητα να είναι μικρότερο το οικολογικό αποτύπωμα των ανθρώπων, αλλά θα αλλάξει και το ίδιο το παράδειγμα. Αυτή η αιμονή με το ΑΕΚΠ και πρέπει να το πω αυτό γιατί στην Ευρώπη ε, σήμερα δεν μπόρεσα να περάσω αυτό το μήνυμα εγώ θεωρώ σχεδόν εγκληματικό να πιστεύουμε ότι μια πολιτική που παράγει ε, κάποια ποσοστά ανεργία στις τάξεις του 27-28% και μιλάμε για ανεργία των νέων πάνω από 50% πάνω από του ε, μισού νέου δηλαδή να είναι άνεργοι, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το υπερασπιστούμε. Θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση των προτεραιοτήτων και οι Ευρωπαίοι πολίτε ζητούν κάτι τέτοιο. Δεν είναι ειδικοί, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το ευρύ κοινό να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό παράδειγμα, αλλά υπάρχουν ε, κάποιοι ειδικοί που παρουσιάζουν τέτοια επιχειρήματα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν κινηθούμε όπως είπε ο Χάνς προς μια αλλαγή παραδείγματος από αυξήσεις ε, οριακές της αποδοτικότητας θα δούμε μια καλή ευκαιρία αλλαγής ε, και εδώ απαντάμε στο γιατί τώρα και γιατί στην Ευρώπη. Γιατί νομίζω και στις δύο περιπτώσεις θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Χάντς, θα ήθελες να απαντήσεις εν συντομία. Ναι, καταρχήν, ε, ναι, είναι παγκόσμια η ατζέντα εδώ δεν έχουμε εναλλακτική. Μπορεί οι άνθρωποι να παραπονιούνται για την παγκόσμια στρατηγική, πόσο αργά προχωρά και την αναποτελεσματικότητά της, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική για μια παγκόσμια πλατφόρμα Βέβαια, έχω ένα θέμα με τους ορισμούς. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στο να ορίσουμε ακριβώς τι είναι μια πράσινη οικονομία. Και θα ξαναθέσω μια ερώτηση σε όλους. Αν σας ρωτούσα εγώ, θα μπορούσατε να μου δώσετε έναν ορισμό ενός σκύλου, θα νομίζετε ότι είμαι τρελός. Καταρχήν και περισσότερο δεν μπορούσατε να το κάνετε αλλά όλοι όταν βλέπουμε ένα σκύλο καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται, είτε αν είναι ένας μεγάλος σκύλος ή είναι ένα μικρό σκύλος, αναγνωρίζουμε ε, τι είναι και ξέρουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πράσινης οικονομίας, ε, διαφέρει αρκετά στη Φιλανδία από τη στην Αιθιοπία. Αλλά σε γενικέ γραμμές ε, θα πρέπει να βγούμε από αυτές τις ατέλειωτες συζητήσεις περιορισμών. Δεν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο, πρέπει να προχωρήσουμε. Επομένω, ε, ξέρω ότι είναι λεπτά ευαίσθητο, λεπτό και ευαίσθητο πολιτικά το θέμα των ορισμών στο Νότο και στις αναδυόνομες οικονομίες. Όμως αυτό που θα είναι μια πράσινη οικονομία θα είναι ουσιαστικά κάτι που θα συνάδει με τις πρακτικές που θα προκύψουν από την εφαρμογή αυτής. Δηλαδή θα δούμε και πώς θα προσαρμοστεί και πώς θα διαμορφωθεί στην Ευρώπη, θα δούμε πού θα μας πάνε οι πρακτικές μας, πόσο μακριά θα μας πάνε και πόσο μεγάλο είναι το κενό και πώς θα το διαχειριστούμε αυτό το κενό και είναι ένας από τους στόχους μας. Έτσι λοιπόν, ως πρώην ακαδημαϊκός, ε, κατανοωμένο ότι είναι σημαντικοί ορισμοί, αλλά δεν νομίζω δε ότι θα πρέπει να μας ε, παραλύσουν ε, οι πολιτικές των ορισμών. κύριος Χάρμπορ. Έχω δύο ακόμα ερωτήσεις ε, που θέλω να θέσω και στη Μόνικα γιατί αναφέρθηκε στο παγκόσμιο. η κυρία Καρολέγκουλη είχε μία ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ναι, καλησπέρα. Η ερώτηση μου αφορά τις θέσεις εργασίας, ε, γιατί στη μετάβαση σε μία πρασίνη οικονομία χρειαζόμαστε περισσότερη αποδοτικότητα και πράσινες τεχνολογίες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερες θέσεις εργασίας. χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας για να τεθούν όλα αυτά σε εφαρμογή σε πρώτο χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ στους πανελίστες για το θέμα αυτό και στον κύριο Μπρονίξ ειδικά. Ο κύριος Γκρέκο είχε μια ενδιαφέρουσα, η κυρία μάλλον, είχε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση να ξεκινήσω από την παρατήρηση. Αν δεν μπορούμε να πετύχουμε την οικονομική ανάπτυξη, τότε θα έχουμε χρηματοοικονομική κρίση και μαζική ανεργία. Η οικονομία δεν μπορεί να μεγενθύνεται για πάντα, εκτός ε, και αν πετύχουμε πλήρη αποσύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης οικονομίας ε, και των πόρων που χρησιμοποιούνται. Και πώς ε, βλέπετε να διαμορφώνεται το μέλλον στο δίλημα αυτό. Καταρχήν, να πω μια φράση σε ό,τι αφορά τις χώρες BRIC. Ενίοτε, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο αν ε, δεν γνωρίζει κάποιος ε, το ιστορικό για να διακόψει το, το, το, τι έχει κάνει κατά τη διάρκεια δεκατιών και να προβεί σε αλλαγή παραδείγματο. Μερικές φορέ είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουμε με το να κατανοήσουμε το σύστημα, την κινητικότητα των σήμων πηγών ενέργεια σε άλλε χώρε. Εμεί αυτό περιμένουμε, παραδείγματο χάρη, ο των πωλήσεων μα. για να ενώσουμε πηγέ ενέργεια, είναι πάρα πολύ ψηλό στι χώρε BRIC και οι επενδύσεις ε, αφορούν περισσότερο τις επενδύσεις ε, στις ε, επικοινωνίες. Έχουν ξεκινήσει όμως σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να μπουν σε ένα εντελώ διαφορετικό τεχνολογικό στάδιο. Τώρα, σε σχέση με τις πράσινες θέσεις εργασίας, αν θέλουμε να διατηρήσουμε το, κοινωνικό, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη, αυτό θα μας κοστίσει και στο μέλλον. Έτσι λοιπόν ο αυτοματισμός θα είναι τμήμα της ανάπτυξης της οικονομίας μας και των εταιριών μας. Από την άλλη πλευρά θα χρειαστούμε θέσεις εργασίας υψηλού με υψηλών προσόντων. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το θέμα του εκπαιδευτικού κενού. Δηλαδή, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, το εκπαιδευτικό σύστημα, τα σχολεία, η κατάρτιση διαβίου θα πρέπει να επικεντρωθούν στο να μην αφήνουν τους ανθρώπους χωρίς εκπαίδευση. Θα ζητήσω από τον Ισμαήλ και τον Χάνς ε, να πούν δύο λόγια για αυτό το θέμα, Χάνς, για το εκπαιδευτικό σύστημα. Νομίζω ότι και το σύστημα της γνώσης, ε, του οποίου αποτελεί τμήμα το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να μπει σε ένα μεταβατικό στάδιο σε στριπτική πλειοψηφία των τμήματων οικονομικών στην Ευρώπη. Το τελευταίο χρόνο υπάρχει ένα μάθημα για τα περιβαλλοντικά οικονομικά που είναι πολύ παράξενο γιατί ε, στο πρώτο μάθημα μακροοικονομικών μαθαίνεις ότι έχεις ε, την εργασία το κεφάλαιο και του φυσικού πόρου για την παραγωγή και τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια περνά στο 80% του χρόνου σου για το κεφάλαιο, 20% στου ανθρώπινους πόρου. και στο τέλο η τελευταία χρονιά γίνεται μια επιλογή για την περιβαλλοντικά οικονομικά, δεν έχει νόημα. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα παράδειγμα για να σας πω ότι το σύστημα γνώσης θα πρέπει επίσης να περάσει μια, μια μετάβαση για τις θέσεις εργασίας. Ε, εδώ μιλάμε για ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των θέσεων εργασίας καταρχήν. Δεν υπάρχει σοβαρή έρευνα που να μπορεί να μας ε, δείξει κατά κάποιο τρόπο ότι ε, αν έχουμε ισχυρή περιβαλλοντική νομοθεσία θα οδηγήσει σε λιγότερη ανταγωνιστικότητα και σε λιγότερες θέσεις εργασίας. Αντίθετα έχουμε την πράσινη οδό για την ανταγωνιστικότητα που εξηγήθηκε ε, πάρα πολύ καλά από κάποιες κορυφαίες σχολές στον κόσμο και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, παγκόσμια προοπτική ανάπτυξη, οι κοινωνικές επιστήμες πολλές φορές λένε ότι η πιο σημαντική ηγεμονία που μπορεί να έχει κανείς στην κοινωνία είναι η ηγεμονία Τη κυρίαρχη σκέψη που δεν σου επιτρέπει να σκεφτείς με διαφορετικούς τρόπους. Και νομίζω για το παράδειγμα της ανάπτυξης, ορισμένους κύκλους, μπορεί να είμαστε κοντά σε μια τέτοια ηγεμονία. Είναι δύσκολο λοιπόν ε, να βγούμε από το παράδειγμα αυτό και να έχουμε ένα διαφορετικό σκεπτικό. Αλλά αν δεχτούμε ότι θα ζούμε καλά μέσα σε συγκεκριμένα όρια, εξορισμού θα πρέπει να το κάνουμε. Είναι τεράστια αυτή η πρόκληση. Είναι κάτι που θα πρέπει να κάνουμε από κοινού και θα υπάρχουν διαμάχες μάχες και συγκρούσεις για το θέμα αυτό αναταραχές αλλά κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει ουσιαστικά να σπάσουμε αυτό το παραδοσιακό παράδειγμα που περιγράφηκε και να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Τρία σημεία ένα για την εκπαίδευση. Πραγματικά είναι ένα θέμα που με συναρπάζει και έχω πολύ ριζοσπαστικές απόψεις. Νομίζω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο το έχουμε εξελίξει τα τελευταία 150 χρόνια και εξελίχθηκε και ένα εντελώ διαφορετικό είδο οικονομία. Ε, στην αρχή λέγαμε στο παιδί όταν ξεκινούσε το σχολείο κάτσε κάτω και κάνει ησυχία και φυσικά ένα παιδί δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο και ζητούσαμε τα παιδιά να κάνουν επαναληπτικά και βαρετά ε, καθήκοντα όταν δεν το κάνουν αυτό, λέμε ότι είναι προβληματικά τα παιδιά και χρειάζονται ειδική προσοχή. Και πολλές φορές, και μερικές φορές και φάρμακα. Αλλά τι κάνουμε τώρα, παράγουμε υπάκους εργαζομένους, γιατί η οικονομία των τελευταίων 100 χρόνων πετούσε κάτι τέτοιο. Όμως ε, τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει τροποποίηση, αλλάζει η οικονομία και ε, τελικά οι μηχανές αντικαθεστούν ε, τους ανθρώπους σε κάποιες θέσεις εργασίας και έχουμε άλλα είδη ε, επαγγελμάτων όπου είναι σημαντικά τα κοινωνικά προσόντα, κοινωνική λεπίδραση και βλέπουμε και αλλαγές αλλού. Νομίζω λοιπόν ότι θα έχουμε μεγάλες αλλαγές και μεταλλάξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα το ερώτημα είναι αν θα συνάδουν με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και με τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία, αλλά όπως και να έχει θα έλθουν αυτές οι αλλαγές. Και το αν θα υπάρχει προσαρμογή έτσι όπως έγινε στο παρελθόν στη βιομηχανική επανάσταση, αυτό θα εξαρτηθεί από τη σοφία των ηγετών μας. Δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω και σχετίζεται με αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε ε, ταπεινοφροσύνη. Α μην ε, προσπαθούμε εδώ να ξοδέψουμε πολύ χρόνο για του ορισμού, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα αλλάξουν αυτοί οι ορισμοί. Και να σας πω τουλάχιστον, λέω την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι ισχύει για όλους εδώ, πριν 20 χρόνια δεν νομίζω ότι κανένας θα μπορούσε να έχει προβλέψει το πλήρη αντίκτυπο του διαδικτύου. Δεν νομίζω ότι 10 χρόνια πριν κανείς δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει τον αντίκτυπο των smartphone και των κινητών ή του facebook. Σας παρακαλώ, το MySpace μέχρι το 2003, το Facebook το 2004, ούτε καν δεκαέτη δεν έχουν έχει κλείσει και είναι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι μέλη. Έτσι, λοιπόν, τώρα αν δω την ικανότητά μου πρόβλεψη 25 χρόνια πριν, μάλλον θα πρέπει να είμαι ταπεινό σε σχέση με το τι θα προβλέψω για τα επόμενα 25 χρόνια με ακρίβεια. Αλλά όπως είπε ο Χάνς, ξέρουμε κατά προσέγγιση τι θέλουμε και το αναγνωρίζουμε όταν το βλέπουμε. Έτσι λοιπόν αν κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι είναι απαιτούμενο και είναι μια κατεύθυνση, δεν είναι συγκεκριμένος ο δικός χάρτης που ακολουθούμε. Και κάτι ακόμη, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο πολλοί άνθρωποι διαισθάνονται και κατανοούν τα θέματα αυτά ακόμη και δεν μπορούν να τα διαρθρώσουν να τα αρθρώσουν, με συγχωρείτε. Χρειάζεται λοιπόν να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ των εμπειρογνωμών και του κενού εν γέννη. Ευχαριστώ πολύ και θα έρθω στην τελευταία ερώτηση. Και ελπίζω να είναι σύντομη η απάντηση. Έρχεται από το Twitter η ερώτηση. Τον Green Amati. που αναφέρεται σε προγράμματα αναδάσωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι πολύ απλή ερώτηση. Είναι σε θέση οι Ευρωπαίοι ηγέτες να ηγηθούν αυτή τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία. Χάνς, αν μπορείτε να μας απαντήσετε αυτήν την ερώτηση αντικειμενικά. Μιας και μου ζητήσετε να σύντομος η απάντηση είναι ορισμένη από αυτούς ναι. Κύριε Κίρχερ, ε, είναι περισσότερο σε θέση να το κάνουν από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια, αλλά παραμένει το ζήτημα της κατανόησης του συστήματος και της ταχύτητας. Δηλαδή όχι μόνο ε, να ορίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον, να προβλέπουμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ε, τα προβλήματα. Κύριος Σερκα... Νομίζω ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα ε, επικοινωνίας με, το, με την κοινή γνώμη, δηλαδή να παρουσιάσουμε στο κοινό, τους πολίτες, ένα όραμα ε, το, στο οποίο να, ε, το οποίο να προσυπογράφει η κοινή γνώμη. Και γι' αυτό βλέπουμε την αύξηση των φασιστικών ή των ακροδεξιών κομμάτων, όχι μόνο στην Ευρώπη, παντού. Είναι λίγο φλού, είναι λίγο δύσκολο να ορίσουμε αυτό το, το ζήτημα. Την κατάσταση σήμερα, απομένως, έχουμε μια κατάσταση όπου όλα είναι ανοιχτά. Και πρέπει να έρθει κάποιο ή μια ομάδα προσώπων που να μας παρουσιάζει ένα όραμα. Την θαυμάζω προσωπικά την Ευρώπη, αλλά σκεφτείτε ότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο, την, την α, λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από τρία χρόνια είχαμε ανθρώπους σαν τον Σούμαν ή τον Μονέ, οι οποίοι κατάφεραν να φανταστούν και να πετύχουν, όχι απλώς να φανταστούν, την ενοποίηση της ε, Ευρώπης. Και φτάσαμε μάλιστα στο σημείο σήμερα η νέα γενιά των Ευρωπαίων πολιτών να μην φαντάζεται καν ότι θα μπορούσε ποτέ να υπάρχει πόλεμο στην Ευρώπη. Δηλαδή κάτι που οι γονεί του ποτέ δεν μπορούσαν να φανταστούν. Η προηγούμενη γενιά δεν μπορούσε καν να φανταστεί την, Ευρώπη, την ε, ειρήνη στην Ευρώπη. Και αυτό το όραμα το παρουσίασαν οι ηγέτες αμέσως μετά τη ε, λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δημιουργήθηκε η ΕΚΑΧ και όλη η υπόλοιπη ευρωπαϊκή θεσμία ε, δεκαετία του 50 και μετά. Λοιπόν, ε, αυτό είναι εντυπωσιακό και άξιζε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι. Ας κοιτάξουμε τους ηγέτες σήμερα. Α κοιτάξουμε του ανθρώπου σήμερα ποιο μπορεί να έρθει και να πει αυτό είναι το όραμά μου για την Ευρώπη και να μην φοβάται που θα τον πούν ονειροπόλο. Ε, αν δεν ήταν ονειροπόλοι πριν 50 χρόνια δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε σήμερα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ που αυθόρμητα χειροκροτήσατε του ομιλητέ, κάτι που σκόπευα να σα ζητήσω να το κάνετε. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να δώσω το λόγο σε όλου και να υποβληθούν όλα τα ερωτήματα αλλά έχετε τη δυνατότητα εδώ στη διεξίωση που θα ακολουθήσει να συζητήσετε με τους ομιλητές. Δίνω τώρα το λόγο στην Αν Κλάβερ, την Σύμβουλο Επιστημονικών Θεμάτων στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις της, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Welcome. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Πρέπει τώρα εγώ να κάνω κάποιες τελικές παρατηρήσεις και γνωρίζω πως ε, περιμένετε να βγείτε έξω να πιείτε το ποτάκι. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Νομίζω πως ο τίτλος της ε, τήσεως αυτής διάλεξης είναι πολύ επιτυχημένο όσον αφορά την βιώσιμη βιωσιμότητα και το πώς μπορεί η οικονομία να βοηθήσει το περιβάλλον. Αλλά είναι μια μεγάλη πρόκληση γιατί τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε πρωτοφανείς αλλαγές και με κάποιον τρόπο, οπωσδήποτε κάποιος της γενιάς μου, έχει δει συνεχή ανάπτυξη και αναμένουμε πως αυτό θα συμβαίνει πάντα, όταν προφανώς δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Και νομίζω πως όλα τα μέλη του πάνελ σήμερα μίλησαν γι' αυτό. Να πω κάτι. Ο Στάινερ του προγράμματος περιβάλλοντος του μας μίλησε για πεπερασμένους πόρους. Και βάση της συζήτησης που είχαμε είναι πως πρέπει να καταλάβουμε πως ζούμε σε έναν πεπερασμένο πλανήτη. Με πεπερασμένους πόρους. Ε, τρία πράγματα όμως δεν είναι πεπερασμένα. Πρώτον, η ηλιοφάνεια. Δεύτερον, βαρύτητα. βαρύτητα θα συνεχίσει να υπάρχει. Και το τρίτο είναι η ανθρώπινη εφευρετικότητα. Με αυτά πρέπει να δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν συνεχίσουμε να ξεχνάμε ή να παραμερίζουμε το στόχο που ακούω συνέχεια, δηλαδή ε, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Για μένα ως ε, βιολόγο ε, αυτό είναι οξύμορο. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, αηφόρο ανάπτυξη, γιατί σε ένα σύστημα που υπάρχει ανάπτυξη κάτι θα αναπτυχθεί, κάτι άλλο θα μειωθεί. Αυτό είναι ο πλανήτης στον οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή. Οπότε ζούμε σε έναν κόσμο όπου εμείς στην Ευρώπη χρησιμοποιούμε τριπλάσιους πόρους ε, από τους άλλους, αναλογικά. Και αυτό σημαίνει πως κάποιος άλλος έχει πολύ λιγότερα. Στην ΔΕ Αμερική πενταπλάσια. Ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το σύστημα. Ο Ισμαήλ Σεραγγελδίνη είπε κάτι που με άγγιξε. Πρέπει δηλαδή να δούμε και την ε, περιβαλλοντική και την κοινωνική βιωσιμότητα. Όχι μόνο δηλαδή να κοιτάμε τους πόρους του πλανήτη, τους φυσικούς πόρους, πρέπει να δούμε και τους ανθρώπινους πόρους. Ε, σας δηλαδή, εμένα, εμείς είμαστε οι ανθρώπινοι πόροι. Και είπε και κάτι άλλο, πως εάν ε, λάβει κανείς τα λάθος μηνύματα, θα χαράξει και λάθος πολιτική. Εμείς στέλνουμε τα α, μηνύματα, οπότε το ερώτημα του εάν υπάρχει κατάλληλη ηγεσία για το μέλλον, η ηγεσία ακούει τη δική μας φωνή. Οπότε πρέπει, δεν μου αρέσει η φράση, πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα στην ηγεσία, να σου πούμε πώς τα απαιτούμε αυτά τα πράγματα και μετά θα τα έχουμε. Για μένα αυτό είναι βασικό. Το άλλο όταν μίλησε η Μόνικα Κίρχνερ. Μου έκανε εντύπωση το παράδειγμα που χρησιμοποίησα για το εάν ε, η αεροπορία είχε κινηθεί τόσο γρήγορα όσο η βιομηχανία των ημιαγωγών. Ένα 767 θα έκανε το γύρο του πλανήτη σε 5 ε, λεπτά με κόστος 500 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν πόσο γρήγορα αναπτύσσονται κάποια πράγματα όπως η ημιαγωγή και όπως μας είπε η Μόνικα αυτό έγινε σε ένα περιβάλλον όπου μάλλον επειδή ήταν ανταγωνιστικό βεβαίως και επικερδές αλλά κατάφερε να έχει αποτελέσματα έχοντας κατά νου και την ε, βιωσιμότητα. Και μετά αυτό το οποίο είπε ο Χάνης Το βασικό για μένα ήταν πως πρέπει να ε, ζήσουμε σε έναν κόσμο χαμηλού άνθρακα, κύκλικό και μίλησε για αντοχή των οικοσυστημάτων. Είναι τίποτα από αυτά προαιρετικό. Για μένα είναι σαφές πως δεν είναι προαιρετικά. Είναι απολύτως αναγκαίο, εάν είναι να στραφούν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι και προσεχώς 9. Η πρόκληση για μένα είναι πάντα. Εάν κάποιος είναι άνετα, ζει σε καλό περιβάλλον και πολλοί από εμά στην Ευρώπη και τον αναπτυγμένο κόσμο γενικώ εκεί βρισκόμαστε, ε, δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα. Γιατί σκεφτόμαστε, ε, εγώ τα έχω αυτά και θέλω να συνεχίσω να τα έχω και αν μου πάρει κάποια, σημαίνει πω η ζωή μου χειροτερεύει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια τεράστια πρόκληση. Γιατί έχουμε μια μοναδική ευκαιρία. Και για εμένα, ως επιστήμονα, είναι κάτι το πολύ συναρπαστικό. Έχουμε την ευκαιρία τώρα, επειδή έχουμε τη γνώση του ότι αυτό το οποίο κάνουμε δεν είναι βιώσιμο, είμαστε σε ένα σημείο καμπής, όπου μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Όχι με το να είμαστε απλά επιστήμονες ή οικονομολόγοι ή πολιτικοί, αυτό μπορεί να γίνει με το να εργαστούμε με τελείως διαφορετικό τρόπο, που θα ενώνει τους πολιτικούς, ε, τους ε, οικονομολόγους, τους επιστήμονες, τους πολίτες και όχι να βρούμε μία λύση, αλλά να έχουμε πολλές επιλογές και δεν συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή γιατί αυτή τη στιγμή κάποιοι λαμβάνουν αποφάσεις αλλά είναι μόνοι τους σε μία αίθουσα και δεν ε, ξέρουν τις διάφορες πιθανότητες. Οπότε χρειάζεται να δούμε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αντί να, είναι, αντί να έχουμε ε, ένα σύστημα έτσι κατά αν θα λέγαμε, πρέπει να έχουμε κατά νου το κοινό καλό. Συμφωνώ λοιπόν με το ότι ναι, να έχουμε μια καλή ζωή. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλές επιλογές για το μέλλον, τόσο συναρπαστικές που μπορούμε να εφεύρουμε, γιατί στην ε, Ευρώπη εφήβραμε το σύγχρονο κόσμο. Και μπορούμε να το ξαναεφεύρουμε. Έχουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε κάποια από τα καλύτερα μυαλά του πλανήτη. Καλύτερη γνώση που δημιουργείται εδώ πέρα. Μπορούμε να το μετατρέψουμε αυτό σε κάτι απτό. Αυτό θα πήγε εσύ, ηγεσία, να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση αυτή όχι μόνο για εμάς, αλλά παγκοσμίω για ένα νέο κόσμο. Που θα είναι νέος και συναρπαστικός. Αυτή η ιδέα της κυκλικής οικονομίας. Πολύ ενδιαφέρουσα. Μπορεί να είναι η ηλικία μου, αλλά στην ηλικία μου εγώ δεν θέλω πλέον να έχω πράγματα γιατί είναι βάρος. Φανταστείτε έναν κόσμο που κανείς δεν ε, έχει τίποτα. Ακούγεται κάπως ουτοπικό, αλλά θα έχουμε πρόσβαση σε πράγματα, χωρίς να είναι στην ιδιοκτησία μας. Η τεχνολογία τώρα μπορεί να δημιουργήσει αυτή την ε, υποδομή. Και θα έχουμε Βεβαίω πράγματα, εμπειρίε χωρίς να έχουμε πράγματα στην ιδιοκτησία μα, θα τα δανειζόμαστε και θα τα δίνουμε μετά. Κάτι το φοβερά συναρπαστικό και μπορούμε να το έχουμε αυτό, εάν αυτό θέλουμε για ένα νέο κόσμο. Και μπορεί έτσι να κινηθεί μια οικονομία. Απλά πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά την οικονομία για να α, την ταιριάξουμε και με αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη. Είχαμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πρέπει να έχουμε αυτή την πρόκληση. Δεν είναι το θέμα κάποιοι, κάποιου επιστήμονα ή οικονομολόγου κάπου. Όλοι πρέπει να στείλουμε τα σωστά μηνύματα για να έχουμε τη σωστή πολιτική για έναν κόσμο καλύτερο όχι μόνο για εμάς στην Ευρώπη αλλά για όλο τον πλανήτη. Όχι τώρα, σε 10, 15, 100 χρόνια. Αυτή είναι η πρόκληση. Και είμαι σίγουρη πως θα συζητήσετε τις λύσεις με το ποτό που θα πιείτε εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Well, thank you very much. Ευχαριστώ. Ο ρόλος μου εδώ δεν είναι να συνοψίσω ότι ο συνάδελφος το έκανε εξαιρετικά. Ο κύριος Ρούμπικ ε, δεν ήταν διαθέσιμος να περευρεθεί εδώ, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, ήλθατε και παρακολουθήσατε όλη τη συζήτηση και θέλω να ευχαριστήσω και όσους συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα από το Twitter και κρατούν ζωντανή τη συζήτηση. Ευχαριστώ και τη γραμματεία της ε, στο ΑΜ και τους ε, συναδέλφους από τη γραμματεία για την οργάνωση αυτής της ετήσιας διάλεξης. Να ευχαριστήσω και τον Malcolm Harbour ε, για το συντονισμό της συζήτησης πολύ ομαλά διεύθυνε την όλη συζήτηση και ευχαριστώ και τον συνάδελφο Όλτριξ Βλάσακ για το εισαγωγικό του για την εισαγωγική του παρέμβαση και τον κύριο Στάινερ από τα Ηνωμένα Έθνη για το μήνυμα μέσω βίντεο. Επίσης ευχαριστώ τους ομιλητές, πραγματικά όλοι εντυπωσιαστήκαμε με το περιεχόμενο των ομιλιών ε, του κυρίου Σεραγγέλτιν, της κυρίας Κίτνερ και του κυρίου Μπρούνιξτ. Σας ευχαριστώ και τους τρεις που παρευρεθήκατε εδώ και δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Και τέλος, την κυρία Γκλόβερ, που δεν είναι κάποια από την απέναντι πλευρά του δρόμου, αλλά συμμερίζεται τις δικές μας αξίες και τις προθέσεις μας για το μέλλον. Ευχαριστώ, Αν, για τα εμπνευστικά σου λόγια και νομίζω ότι μας βοήθησες να λύσουμε το ξύμερο της βιώσιμης ανάπτυξης με τα τελικά σου λόγια. Και αν ε, δεν ε, επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό μέσω του κοκτέιλ, της δεξίωσης που ακολουθεί, ας γίνουμε κάπως πιο αισιόδοξοι. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Σας ευχαριστώ. Thank you, Malcolm.